Ερωτήσεις προς την Επιτροπή δεν έχουμε λάβει. Ως προς το χρόνο ερωτήσεων, το θέμα αυτό για την ημερησία μας και αφού δεν υπάρχουν τέτοιες ερωτήσεις, μπορώ να προχωρήσω ευθύς αμέσως στο σχέδιο εκθέσεως που αφορά τις ε, επιπτώσεις της παγκόσμιας δημοσιονομικής, χρηματοπιστωτικής συγγνώμη, και οικονομικής κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και την ε, αναπτυξιακή συνεργασία, με ανταλλαγή απόψεων με τον εισηγητή μας κύριο Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σε μια προηγούμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας είχα την ευκαιρία να υποβάλω τις γενικές γραμμές της έκθεσής μου. Σήμερα έχω το σχέδιο έκθεσης Έχει κλείσει το μικρόφωνο του ομιλητή, δεν τον ακούμε. Έλεγα λοιπόν ότι σε μια προηγούμενη συνεδρίασή μα ε, μου είχε δοθεί ευκαιρία να σα παρουσιάσω τι γενικέ κατευθυντήριε γραμμέ τη έκθεσή μου. Και ότι σήμερα έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω το σχέδιο έκθεσης όσον αφορά τις συνέπειες από την οικονομική και δημοσιονομική κρίση στις υπονάπτυξη χώρες. Θέλω να ξεκινήσω με την ε, λογική που ακολουθώ στην έκθεσή μου. Σήμερα αντιμετωπίζουμε μια κρίση ανάπτυξης η οποία είναι συνέπεια της οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης η οποία ξεκίνησε στα τέλη του 2007. Όμως, Πέρα από αυτή τη διαπίστωση, η έκθεση υπογραμμίζει επίσης ότι αυτό το οποίο ήταν σε κρίση ήδη πριν από το 2007 ήταν η ίδια η αναπτυξιακή πολιτική. Και γιατί ήταν σε κρίση η αναπτυξιακή μας πολιτική. Γιατί πέρα από το γεγονός ότι οι ανάπτυξη χώρες αναπτύσσονταν, παρά μάλλον αυτό το γεγονός και παρά το γεγονός ότι η αναπτυξιακή βοήθεια αυξάνεται, και παρά τα σημαντικά επιτεύγματα που έχουν πετύχει πολλές χώρες, παρόλα αυτά, αντί να πλησιάζουμε στους στόχους της χιλιετηρίδας, απομακρυνόμασταν από αυτούς. Δηλαδή, το έτος 2007, πριν να ξεκινήσει η κρίση, ήδη είχαμε απομακρυθεί από τους στόχους της χιλιετίας, αντί να βρεθούμε πιο κοντά σε αυτούς όπως θέλαμε. Συνεπώς υπάρχει εδώ πέρα μία διπλή προοπτική στην έκθεση αυτή. Αφενός μιλάμε για τα μέτρα. Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε για να λυθούν προβλήματα τα οποία απορρέουν από την κρίση, άμεσα μέτρα. Και κατά δεύτερον, πρέπει να δούμε τι καινοτομίε χρειαζόμαστε προκειμένου να τροποποιήσουμε την πολιτική μας ανάπτυξης, προκειμένου μέσω πρόθεσμα να ε, φέρουμε σε πέρας τις υποχρεώσεις μας με την λήξη της οικονομικής ε, κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Πώς να αντιμετωπιστούν λοιπόν μέσω πρόθεσμα τα αναπτυξιακά ζητήματα. Για να γίνει αυτό απαιτούνται, απαιτείται καινοτομία. Απαιτούνται νέες πηγές χρηματοδότησης επίσης για την ανάπτυξη απαιτείται πιο αποτελεσματική διαχείριση των αναπτυξιακών πολιτικών και απαιτείται μια πιο δημοκρατική εκπροσώπηση στα διάφορα δημοσιονομικά διεθνή όργανα, ώστε οι υπονάπτυξη χώρες να έχουν περισσότερα περιθώρια στη διάθεσή τους. Χρειάζεται επίσης μεγαλύτερη υπευθυνότητα, μεγαλύτερη αυτονομία των χωρών που λαμβάνουν αναπτυξιακή βοήθεια. Χρειάζεται επίσης μεγαλύτερη παρέμβαση από πλευράς της κοινωνίας των πολιτών και χρειάζεται μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Πρέπει δηλαδή να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες και από την κοινωνία και από τον ιδιωτικό τομέα και από το δημόσιο τομέα που να προσφέρουν νέο δυναμισμό στις αναπτυξιακές μας πολιτικές. Η έκθεση λοιπόν που σας παρουσιάζω σήμερα περιλαμβάνει μέτρα άμεσου χαρακτήρα και περιλαμβάνει επίσης και προτάσεις μεταρρύθμισης για αργότερα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα ώστε οι καινοτομίες αυτές οι οποίες αναφέρθηκαν να συμπεριληφθούν στην αναπτυξιακή μας πολιτική. Γνωρίζετε, γνωρίζει και η Επιτροπή και το Συμβούλιο και οι Ευρωβουλευτές. Όλοι όσοι βρίσκονται εδώ σήμερα το γνωρίζουν ότι υπάρχουν επίγοντα προβλήματα τα οποία πρέπει να λυθούν εξαιτία της κρίσης προβλήματα. Είμαστε σε μια κατάσταση μείωση της ανάπτυξη, μείωση της τιμή των πρώτων υλών Οι χώρες δηλαδή που εξάγουν πρώτες ύλες βλέπουν ότι μειώνονται οι τιμές τους και συνεπώς οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν επιπλέον και εμπορικούς περιορισμούς και προστατευτισμό από άλλες χώρες με προβλήματα αξεπέραστα. Παίρνουν βάσματα από τους μετανάστες τους βέβαια, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα έσοδα των χωρών αυτών, αλλά παρόλα αυτά ε, συγκεντρώνουν και συσσωρεύουν μεγαλύτερο χρέος και παίρνουν έτσι και λιγότερη αναπτυξιακή ενίσχυση. Όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας και να τα αντιμετωπίσουμε. Και γρήγορα μάλιστα. Όπως είπα όμως και πριν, Υπάρχει και μεσοπρόθεσμα ε, κάτι που μπορούμε να κάνουμε και είναι η καινοτομία στην οποία αναφέρθηκα πριν. Η έκθεσή μου λοιπόν περιλαμβάνει, την έχετε εξάλλου όλοι νομίζω στη διάθεσή σας και σε όλες τις γλώσσες. Περιλαμβάνει κάποιες προτάσεις και θα αναφερθώ σε μερικές από αυτές γρήγορα. Γιατί δεν αξίζει τον κόπο να μπω σε λεπτομέρειες προτιμάω να ακούσω μετά την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τους συναδέλφους τι έχουν να μου πούνε. Λοιπόν, η έκθεσή μου ζητάει ενίσχυση των ε, στόχων της χιλιετίας. Δηλαδή, να κάνουμε μεγαλύτερη προσπάθεια για να πετύχουμε αυτούς τους στόχους το 2010. Το φθινόπωρο του 2010 στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενική Συνέλευση θα πρέπει να υπάρξει ε, μια, ένας απολογισμός για το σε τι βαθμό έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της χιλιετίας. Και πρέπει συνεπώς να αναλάβουμε τη δέσμευση ότι το 2015 θα έχουμε κάνει αυτά τα οποία προτείναμε το 2000. Δεν είναι δυνατόν να πούμε «Α, δεν τα καταφέραμε, δεν πειράζει» να σταματήσουμε τις προσπάθειες όσο δεν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι Τη χιλιετία έχουμε πέντε χρόνια ακόμα μπροστά μας. Άρα πρέπει να παλέψουμε για να τα καταφέρουμε. Η έκθεσή μου επίσης θέλει οι χώρε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίσης να φέρουν σε πέρα τι υποχρεώσει τους για το 0,56% του ΑΕΠ του 2000 και 0,7% το 2015. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να φροντίσουμε να καλύψουμε τους στόχους που εμείς ήδη βάλαμε και να αποτελέσουμε εμείς παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο, για τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου ή για άλλους διεθνείς οργανισμούς. Η έκθεσή μου επίσης μιλάει για την αναγκαιότητα που υπάρχει να βρούμε επιπλέον πηγές χρηματοδότησης. Το είπα αυτό και πριν. Επίσης υπογραμμίζει ότι πρέπει να πετύσουμε από τα, τους διεθνείς ε, δημοσιονομικούς οργανισμούς, την Παγκόσμια Τράπεζη, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, να δανείσουν γρήγορα στις αναπτυσσόμενες χώρες όχι να κάνουν υποσχέσεις για δάνεια που έχουν γίνει πολλές τα τελευταία δύο χρόνια χωρίς όμως τα δάνεια να έχουν φτάσει ποτέ στον προορισμό τους. Πρέπει να προσέξουμε πολύ αυτό γιατί αυτά τα δάνεια ή υποσχέσεις δανείων καλύτερα χρεώνουν ακόμα περισσότερο τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο στην επίτευξη των στόχων τους. Τώρα για τις νέες πηγές χρηματοδότησης. Η έκθεση μιλάει για την εισαγωγή ενός φόρου όσον αφορά τις διεθνείς οικονομικές συναλλαγές. Και όχι μόνο προκειμένου να διατηρηθεί το οικονομικό σύστημα ή για να μπορέσουμε να πάρουμε πίσω τα χρήματα τα οποία δώσαμε στις τράπεζες για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που είχαν. Ένα μέρος ναι, αλλά πάνω απ' όλα για να πετύχουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό αναπτυξιακής βοήθειας. Προτείνω επίσης να υπάρξει ένα μνημόνιο όσον αφορά την πληρωμή του χρέου. Οι αναπτυσσόμενες χώρε, δηλαδή, οι οποίες σήμερα χρεώνονται ακόμα περισσότερο εξαιτία των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν, να έχουν ένα μνημόνιο, τριετές, προκειμένου να επιστρέψουν τα χρέη τους. Επίσης, προτείνω και την εισαγωγή ε, φόρου περιβαλλοντικού ε, φόροι δηλαδή στις μεταφορές για παράδειγμα, γιατί είναι ορισμένες χώρες οι οποίες σε θελοντική βάση θέλουν να το κάνουν. Στο μέλλον θα αποτελέσει ένα πραγματικό μέσο αντιμετώπισης των ε, περιβαλλοντικών ε, προβλημάτων. Επίσης, η έκθεσή μου προτείνει οι χώρες ε, εκείνες από τις οποίες ε, φεύγουν εμβάσματα και πάνε στις αναπτυξιακές χώρες να αφαιρεθεί το ποσό από τους μετανάστες αυτούς των χρημάτων που πρέπει να πληρώνουν για να στέλνουν εμβάσματα στις χώρες τους. Και οι χώρες οι οποίες παίρνουν τα εμβάσματα να μην ε, βάζουν φόρο στα χρήματα αυτά που φτάνουν στη χώρα απ' έξω στην ε, Λάκυλα το 2008 ε, συζητήθηκε αυτό μείωση δηλαδή του φόρου που ε, μπαίνουν στα εμβάσματα αυτά. Η έκθεση επίσης υπογραμμίζει όλος ιδιαιτέρως τις πρωτοβουλίες ιδιωτικού δημοσίου τομέα διότι θεωρώ ότι η ιδιωτική πρωτοβουλία από τις ιδιωτικές δηλαδή επιχειρήσεις είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό μέσο προκειμένου όχι να έχουμε αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά επενδύσεις στις ε, υποανάπτυξη χώρες. Και άρα θα υπάρξει έτσι και μεταφορά τεχνολογίας, ε, μεταφορά know-how, ώστε αυτό που τώρα λέμε aid for trade, βοήθεια δηλαδή για μέσω του εμπορίου θα γίνει πολύ περισσότερο πραγματικότητα στο μέλλον. Προτείνει επίσης η έκθεσή μου κάτι για το γύρο της ε, Ντόχα. Να επιτευχθεί εκεί συμφωνία που να μην είναι περιοριστική για το εμπόριο γενικά. Ούτε να είναι περιοριστική όσον αφορά ειδικά το εμπόριο των ε, υποανάπτυξη χωρών οι συμφωνίες οικονομικής ε, σχέσης να αποτελέσουν ένα μέσο ανάπτυξης, κάτι το οποίο βέβαια απαιτεί γρήγορα διαπραγματεύσεις μέχρι το 2010. Η έκθεσή μου επίσης ε, μιλάει κατά των οικονομικών παραδείσων. Είναι και αυτό ένα θέμα που έχει βάλει σαν προτεραιότητά της η Ισπανική Προεδρία που ξεκινάει μάλιστα σε δύο εβδομάδες. Όπως και άλλα θεσμικά όργανα, έτσι και εμείς θέλουμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να βάλουν πιο αυστηρά κριτήρια, να είναι πιο απαιτητικοί απέναντι στη διαφάνεια των ε, δημοσιονομικών αυτών παραδείσεων Προς το παρόν, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η ΟΣΑ, δεν βάζουν πολύ αυστηρά κριτήρια. Οπότε και ο ΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων πρέπει να αναθεωρήσουν τα κριτηριά τους και να είναι πιο αυστηρά όσον αφορά την διαφάνεια των ε, δημοσιονομικών συναλλαγών. Πρέπει να είναι πιο αυστηρά τα κριτήρια που έχουν να κάνουν με τους οικονομικούς παραδείσους, δημοσιονομικούς παραδείσους. Λέει επίσης η έκθεσή μου ότι προοδευτικά, σιγά σιγά, αλλά σταθερά, οι πολυεθνικές Επίσης, να αποκτήσουν μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τις συναλλαγές τους. Πολύ συγκεκριμένα, κατά περίπτωση και όχι έτσι γενικά, ώστε να αποτελούν κάτι που ξεφεύγει από τον έλεγχό μας. Συγχρόνως ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να δρά βάσει αυτών των κριτηρίων. Θέλω επίση και μέτρα κατά της διαφθορά. Περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τη φορολογία. Αυτό το σύνολο δράσεων που σας ανέφερα έχει βέβαια μια λογική. Έτσι. Δεν πρόκειται για μια συσσόρευση μέτρων. Πρόκειται για δράσεις, όπως είπα και στην αρχή, που πρέπει να αναλυφθούν μέσα στο 2010 για τα επίγοντα ζητήματα και υπάρχουν και δράσεις οι οποίες πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή αργότερα ή σιγά σιγά προκειμένου να ε, καλύψουμε τους στόχους που έχουμε βάλει. Θα ολοκληρώσω με το εξή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αναπτυξιακής πολιτικής. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε μία θέση ε, από την οποία θα αποτελούμε παράδειγμα καλών πρακτικών. Σίγουρα υπάρχει και μια ηθική διάσταση σε όλα αυτά. Πάντως πρέπει να είμαστε παράδειγμα για άλλες χώρες με τις καλές πρακτικές που εφαρμόζουμε ώστε να συμμετάσχουν όλο και περισσότεροι στην αναπτυξιακή πολιτική. Τέλος, με την έκθεσή μου θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα εμείς, η Αναπτυξιακή Επιτροπή, πρέπει να είμαστε στην πρώτη γραμμή και να παρασύρουμε και άλλους μαζί μας υπέρ της αναπτυξιακής βοήθειας και αργότερα να μπορέσουμε να ελέγξουμε κατά πόσο οι καινοτομίε αυτές που προτείνουμε τίθενται σε εφαρμογή ή όχι. Ο εισηγητή είμαι στη διάθεσή σας, είμαι ανοιχτό για ό,τι παρατηρήσεις, σχόλια, ε, προτάσεις Καινοτομίε, έχετε να προτείνετε. Περιμένω και τροπολογίες από εσά. Ό,τι τροπολογίες έχετε, ευχαριστώ. Υπόσχομαι ότι θα τις μελετήσω και θα προσπαθήσω να είμαι όσο γίνεται πιο ελαστικός για να συμπεριλάβω όσο γίνεται περισσότερες από τις τροπολογίες σας στην έκθεσή μου. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Mr. Um... Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Ρουτιχώσνο, να μας πει δύο λόγια. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Επιτροπή θεωρεί ευπρόσδεκτη αυτή την έκθεση. Κύριο κύριε Σαλόμ, υποστηρίζουμε όλα όσα είπε ο κύριος Βουλευτής και ιδιαιτέρως θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμιστεί το γεγονό ότι όντω η χρηματοπιστωτική και η οικονομική κρίση θα έχει πολύ πιο ισχυρές τραγικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη των ε, αναπτυσσομένων χωρών, στους λαούς των αναπτυσσομένων χωρών και υπάρχει ασφαλώς διασύνδεση μεταξύ της κρίσης και της κατάστασης αυτών των οικονομιών. Θα επανέλθω όμω. Όπως είπε ο κύριος Γερόνος Σαλόμ, θα θυμάστε κι εσείς ότι στην αρχή του έτους όταν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη πρότειναν ε, με ζήλο ε, σχέδια διάσωσης ή ανάκαμψης, όπως άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στις 8 Απριλίου πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα πρόγραμμα διάσωσης για τα κράτη της ε, ΑΚΕ όταν κανείς άλλος δεν είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό ακόμη και όταν ακόμη και η ομάδα των 20, το G20, είχε ασχοληθεί μόνο με τι ανεπτυγμένε και όχι με τι αναπτυσσόμενε χώρε. Πράγμα το οποίο αργότερα άλλαξε. Αλλά τη στιγμή που η Επιτροπή έκανε την ανακοίνωσή τη, ήμασταν λίγο πολύ οι μόνοι οι οποίοι έκρουαν τον κόδωνα του κινδύνου τόσο ενωρί ω προ τη σοβαρότητα των ε, επιπτώσεων αυτής της κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες. Έχουμε μάλιστα εκείνη την εποχή καταθέσαμε ένα κατάλογο ολόκληρο μέτρων που δεν διαφέρει από τα όσα μας ε, εξέθεσε ο εισηγητής. Οπότε θα αυτές σε λεπτομέρειες. Πλην όμως θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι με την ανακοίνωσή μας, στην ανακοίνωσή μας το Συμβούλιο αντέδρασε ως εξή. Ε, καλώς όρισε την ανακοίνωση, θεώρησε ευπρόσδετα όσα λέμε, αλλά δήλωσε σαφώς ότι δεν πρόκειται να διαθέσει ούτε μία δεκάρα, ούτε ένα λεπτό του ευρώ ε, σε ένα νέο πρόγραμμα διάσωσης. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η πίεση προς το Συμβούλιο για την ε, διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου στήριξης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προς τα κράτη αυτά. Και επίσης, ναι, μπορεί τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να έχουν ε, δημιουργήσει ένα νέο σύνολο μέσων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Τα περισσότερα από αυτά τα μέσα δεν ε, αφορούν τις ελάχιστα ανεπτυγμένες χώρες. Για χώρες μέσου εισοδήματος και κάποιες από τις λιγότερο ανεπτυγμένες μπορεί να είναι χρήσιμα, αλλά πολλές από τις χώρες αυτές δεν μπορούν να τα αξιοποιήσουν αυτά τα μέσα ή αν τα αξιοποιήσουν, απλώς τα αξιοποιούν με κόστος, με τίμημα, την αύξηση του εξωτερικού του χρέου, πράγμα το οποίο βεβαίω δεν μπορούμε να ζητούμε από αυτές, όταν ύστερα από 10 χρόνια σκληρών προσπαθειών κατάφεραν να μειώσουν μαζί μα το χρέος τους σε αυτές οι αναπτυσσόμενες χώρες. Γι' αυτό η Επιτροπή προτείνει να υποστηριχθεί μια σειρά προγραμμάτων, σχεδίων που έχουν αναπτυχθεί μαζί με τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ως προς την αφορία του χρέους ή την παρακολούθηση, την επιτήρηση του χρέους, πράγμα το οποίο θα σήμαινε ότι δεν θα χρειαστεί μέσα σε μερικά χρόνια να ξαναρχίσει ένας νέος γύρος ε, προσπαθειών για ανακούφιση του χρέους αυτών των χωρών. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον εισηγητή για την αναφορά του στην πρόταση της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός νέου μέσου, αυτό που ονομάζουμε Vulnerability Flex, ευέλικτο μέσο ευαλωσιμότητας, πράγμα το οποίο ε, αναπτύξαμε πρέπει να σας πω σε στενή συνεργασία με τους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με πολύ καλή ε, συμπληρωματικότητα στις προσπάθειές μας γιατί ενώ τα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προτείνουν νέα δάνεια εμείς προτείνουμε ε, χορηγίες, δωρεές δηλαδή. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και έχουμε μπορέσει πιστεύω να συμφωνήσουμε ως προς τον κατάλογο εκείνων των κρατών που χρειάζονται περισσότερο τα ποσά αυτά των δωρεών και για να ευλογήσω και τα γένια μου πρέπει να σας πω ότι λίγους μόνο μήνες χρειαστήκαμε για να δημιουργήσουμε ένα νέο μέσο και για να κινητοποιήσουμε να κατανείμουμε και να διαθέσουμε τους σπόρους από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης ε, μέσα σε μερικούς μήνες όπως είπα. Είμαστε ο μόνος χορηγός που μπόρεσε να ανταποκριθεί αποτελεσματικά με τρόπο κύκλικό και τη στιγμή κατά την οποία ε, η ε, συνθήκες ήταν οι χειρότερες και οι ανάγκες ήταν οι υψηλότερες. Θα ήθελα επομένω να επισημάνω ότι σε μερικέ ημέρε θα υπάρξει μια, ένα ανακοινωθέν τύπου που ήδη θα ενημερώνει για τι χώρε οι οποίε θα μπορέσουν να υποφεληθούν από αυτού του μέσου, του Vulnerability Flex και βέβαια θα συνεχίσουμε και το 2010 την υποστήριξη. Επίση θα ήθελα να, να υπογραμμίσω τα όσα είπε ο εισηγητή για τα φορολογικά συστήματα στι αναπτυσσόμενε χώρε, γιατί είχαμε μια μεγάλη διάσκεψη εδώ ακόμη χτες ε, με την Εύα Ζολή στην αίθουσα που βρισκόμαστε τώρα ε, για την σημασία ε, του να, αποδοθεί, του να δοθεί έμφαση στα φορολογικά συστήματα στις αναπτυσσόμενες χώρες έτσι ώστε να μπορούν τα αναπτυσσόμενα κράτη να συλλέγουν τους πόρους τους, να έχουν ιδίους πόρους και να δρουν αυτό δύναμα. Αυτό είναι ανάγκη, ε, είναι ε, συναφές με την ανάγκη της ίδιας επιβίωσης των κρατών αυτών και δεν αφορά αποκλειστικά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι σε λίγου μήνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει τις προτάσεις ε, εκθέσεων για την επίτευξη των στόχων ODA που θα συνδυάσουμε εφέτος και με μια ανακοίνωση ως προς τη φορολογία σε σχέση με την ανάπτυξη, το λεγόμενο ε, εαρινό πακέτο εκθέσεων, στο οποίο αναφέρονται, αναφέρονται τα ποσοστά επίτευξης των στόχων του Μοντερέι. Με τη νέα αυτή λοιπόν ε, πρόταση καταθέτουμε ε, ιδέες με ύψιστη προτεραιότητα, με συγκεκριμένα μέτρα που θα αφορούν και τη δική μας αναπτυξιακή συνεργασία με τα αναπτυσσόμενα κράτη. Και για να καταλήξω, συμφωνούμε πλήρως με την έκθεση αυτή. Σε ένα μόνο μικρό σημείο θα θέλαμε να ζητήσουμε τη διόρθωση ότι αφού ε, κινητοποιούμε ποσά που δεν έχουν κατανεμηθεί ακόμη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης, δεν πρόκειται για προκαταβολή, η οποία ενδεχομένω θα προκαλέσει προβλήματα αργότερα. Πρόκειται για χρήση κονδυλίων που ούτω ή άλλω θα διέθετε το ADF κατά τη διάρκεια τη λειτουργία του. Και πιστεύουμε ότι είναι τώρα η στιγμή να κινητοποιηθούν, να διατεθούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη επίσης πρέπει να σημειώσω ότι είναι de facto το μόνο μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει αποθεματικό. Τα άλλα δεν μπορούν να διαθέσουν από τα αποθεματικά τους κονδύλια για να αντιμετωπίσουν μια έκτακτη κρίση. Πράγμα το οποίο είναι και τροφή για σκέψη για το μέλλον, ίσως δηλαδή για τα ε, μέσα ανάπτυξης, τα αναπτυξιακά μέσα που θα έχουμε στο μέλλον. Μόνο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη μπορούμε να στηριχθούμε και τα υπόλοιπα δεν θα είναι εξίσου χρήσιμα για μια ε, χώρα σε κατάσταση κρίσης. Η μόνη δηλαδή πρόσθετη χρηματοδότηση που μπορεί να εξασφαλιστεί, όσο χρήσιμα και τα άλλα μέσα χρηματοδότηση για την ανάπτυξη, ε, η μόνη όμως αξιόπιστη πηγή χρηματοδότηση που μπορεί να βρεθεί σε περίπτωση κρίση είναι το EDF. Ο Πρόεδρος, δηλαδή, εάν κατάλαβα καλά, μπορούν να αξιοποιήσουν, ε, μπορούν να υποφεληθούν αυτό που αποθεματικού τα κράτη και... Και θεωρείτε ότι σε σχέση με τον πληθυσμό και τις ε, γραμμές LA εφέτος στον προπολογισμό υπάρχουν κράτη τα οποία δεν θα μπορέσουν να υποφεληθούν, Λατινική Αμερική. Και το DCI και το ENPI, τα άλλα αναπτυξιακά μέσα δηλαδή, έχουν ήδη προγραμματίσει την ε, κατανομή των ποσό Δεν έχουν μείνει δηλαδή αδιάθετα ποσά και ως εκ τούτου δεν υπάρχει περαιτέρω δυνατότητα διάθεσης κονδυλίων. Είναι πολύ περιορισμένο το πεδίο που θα είχαμε για προκαταβολή, front loading, που όμως θα σήμαινε ότι υποθηκεύουμε τα επόμενα χρόνια. Για δε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης είχαμε προβλέψει κάποια σημαντικά ποσά στο αποθεματικό που δεν είχαν διατεθεί, άρα μπορούμε να τα ε, χρησιμοποιήσουμε, αλλά βέβαια και πάλι πρέπει να ξέρουμε ότι αν σε δύο χρόνια εμφανιστεί μια χειρότερη κρίση, πάλι θα είναι πολύ περιορισμένο το παθηματικό μα. Αυτό πρέπει να έχουμε υπόψη. Και με αυτό να λάβουμε τι αποφάσει που θα λάβουμε σε αυτή τη στιγμή. Και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη δηλαδή, ε, περιορίζουμε λίγο πολύ τι δυνατότητε ανταπόκριση σε μια κρίση που ενδεχομένω εμφανιστεί σε δύο χρόνια. Ο Πρόεδρο, κύριε Διευθυντά, χώρε όπω το Μπαγκλαντέ, Μαλδίβε, και άλλες χώρες της Ασίας. Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι κινδυνεύουν να υποστούν πολύ σημαντικές ε, ε, πολύ, προσημα... πολύ σημαντική επιβάρυνση ως προς την προσαρμογή του στην κλιματική αλλαγή ε, προτάσεις οι οποίες άλλωστε θα κοστούν σε λίγο στην Επιτροπή μας 30 εκατομμύρια ανθρώπων θα χρειαστεί να βρουν άλλο μέρος για να χτίσουν το σπίτι τους, για να κατοικήσουν σε λίγο λόγω των κλιματικών αλλαγών. Δεν μπορούμε λοιπόν να περιοριζόμαστε μόνο στην Αφρική και την ΑΚΕ για την προσφορά υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ ως Ασιάτης ο ίδιος. Πρέπει να πω ότι έχει τεράστιες ανάγκες η Ασιατική Ήπειρος. Πρόεδρε, δεν έχω πραγματική απάντηση στο ερώτημά σας. Η πραγματική απάντηση Ελπίζω να δοθεί από την Κοπενχάγη. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι ειδικά για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης αλλά και για τα υπόλοιπα μέσα και εργαλεία που έχουμε προσπαθούμε να δούμε πώς θα επαναπροσανατολίσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια λόγω της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της. Παραδείγματος χάρη, είμαστε σε μια φάση όπου κάνουμε ενδιάμεση αναθεώρηση όλων των ε, εγγράφων ε, των, της στρατηγικής αναχώρα και δίνουμε εντολές ε, στις αντιπροσωπείες και στις ε, χώρες γιατί στέλνουμε επιστολές από τους επιτρόπους στις αντιπροσωπείες και στις χώρες εταίρους να εξετάσουν στις ενδιάμεσες εκθέσεις τους τι δυνατότητες υπάρχουν για να επαναπροσανατολίσουμε την αναπτυξιακή βοήθεια, αν γίνεται μεταξύ άλλων και για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. Επομένως, στην αναπτυξιακή μας βοήθεια θα πρέπει να ψάξουμε ήδη τρόπους ούτως ώστε να καταπολεμήσουμε την ε, κλιματική αλλαγή με αλλαγή προτεραιοτήτων. Αυτή ξέρω ότι είναι μία μερική απάντηση, αλλά χρειάζεται να δοθεί και αυτή η απάντηση. Για αυτό το σημείο, λέει ο Πρόεδρος. Πριν από δύο μέρες συναντήθηκα ε, με πολλούς ανθρώπους ε, όπου συζητήσαμε την κλιματική αλλαγή και την απώλεια υδάτων ε, στη Σομαλία. Η UNDP μου είπε ότι η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να αυξήσει την ανάπτυξη. Επομένως τα πράγματα δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, είναι και το ένα και το άλλο. Ο κύριος Κάσμαν. Ευχαριστώ πρόεδρε. Παρεμβαίνω για να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε, για την συνολική και σφαιρική προσέγγιση που έχει για αυτό το εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Με μεγάλη χαρά κοίταξα ότι είδα ότι έχει τα φορολογικά καθεστώτα συμπεριλάβει στην έκθεσή του και το θέμα της φοροαποφυγής και διαφυγής και καλωσορίζω τη σημασία που θα δώσει η Ισπανική Προεδρία σε αυτά τα θέματα. Επίσης, ε, ασχολείται και με το θέμα των εμβασμάτων. Ξέρουμε ότι τα εμβάσματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες ξεπερνούν κατά πολύ την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Και αυτό είναι περίεργο. Ε, γιατί οι ενδιάμεσοι πραγματικά ε, βγάζουν πολλά λεφτά και οι χώρες αυτές στερούνται έτσι πόρων. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ηνωμένου Βασιλείου, ούτω ώστε ε, να μειώσουμε το κόστος της αποστολής εμβασμάτων. Επίσης, δόθηκαν πάρα πολλά λεφτά στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή. Το 1,6 ή 1,7% από αυτά μόνο έφτασε σε αναπτυσσόμενες χώρες, από αυτά τα λεφτά. Το 86% πήγε στις λεγόμενες αναβιώμενες δημοκρατίες και αναδυόμενες χώρες. Αυτό είναι ενδιαφέρον όταν βλέπουμε τα προβλήματα που έχουν χώρες μεσαίου εισοδήματος όπως λέγονται, που πριν ήταν αναπτυσσόμενες χώρες. Θα το ξανααναφέρω αυτό. Μόλις γύρισα από την αποστολή στην Ποτσουάνα. Ε, βλέπουμε εκεί μια χώρα όπου την κατατάσσουμε στην, ε, στις χώρες μεσαίου εισοδήματος. Έχει πρόσβαση στα προγράμματα χρηματοδότηση από τους δωρητές, αλλά η πρόσβαση αυτή έχει μειωθεί τώρα. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν τις ειδικέ ανάγκες και τα ειδικά προβλήματα που έχουν ορισμένες χώρες. Ε, να ξαναδούμε μια χώρα όπως η Μποτσουάνα και άλλες ε, χώρες τέτοιου, που έχουν τέτοια προβλήματα. Να δούμε επίσης ε, τι βοήθεια δίνει το κράτος σε ανθρώπους που είναι φορείς του AIDS ή είναι άρρωστοι από AIDS. οι, μη, λιγότερο αναπτυσσόμενες χώρες, αναπτυγμένες χώρες έχουν επηρεαστεί και οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν επηρεαστεί. Αλλά ξεχνάμε, ξεχνάμε κάπου τις ε, ενδιάμεσες χώρες, τις ε, χώρες δηλαδή μεσαίου εισοδήματος. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι είναι μεσαίου εισοδήματος. Είναι μια αντίληψη αυτή. Τώρα το θέμα του ποσοστού που θα δώσουν τα κράτη-μέλη για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ε, σίγουρα δεν τα πάμε καλά. Και το επιχείρημα ότι επειδή εμείς έχουμε πρόβλημα, α, δεν πρέπει και, οι άλλοι να, πρέπει και άλλοι να έχουν πρόβλημα, αυτό δεν είναι σωστό. Υποφέρουμε εμείς, άρα θα υποφέρουν και οι άλλοι. Ε, μιλάμε για το 0,7% του ΑΕΠ, ε, τα 100 του ΑΕΠ. Εγώ, κοιτάξτε, είμαι άσχετος από μαθηματικά, είμαι άσχετος από οικονομικά. Αλλά αν κάποιος ε, έρθει σε μένα, μπορώ να τα, πω έτσι πολύ, να τα πούμε πολύ σύντομα αυτά τα θέματα, ε, είτε στο μπάρ είτε στο γραφείο μου. Επίσης, ε, χαιρετίζω την προσέγγιση του εισηγητή. Οι δραματικές επιπτώσεις δεν πρόκειται να γίνουν αισθητέ. Είναι ήδη αισθητέ. Και επομένως οι συστάσεις που προκύπτουν από την έκθεσή σας και από την ε, δέσμευση που έχει αναλάβει η Κομισιόν είναι ευπρόσδεκτες. Να επανέλθω στην ε, ιδεολογία του Μάρξ για τα αποθέματα. Πρέπει να κρατήσουμε τα αποθέματα. Τα χρειαζόμαστε. Τέλος πάντων, κάπου πρέπει να διοχετευτούν αυτά τα αποθέματα και ενδεχομένως να πετύσουμε από τα κράτη-μέλη να δώσουν, να, να, κάπως αυτά τα αποθέματα. Κάθε χρόνο το κάνουμε ετήσια. Θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να το κάνουμε και σε επίπεδο 27, ε, να δράσουμε όμως ενωμένα. Αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να ονομαζόμαστε ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση του Γκράουτσο Μάρξ. Ή θα μπορούσαμε μάλλον να ονομαζόμαστε. Μ' άρεσε η έκθεση. Χαιρετίζω τον εισηγητή ε, και το, για τη δουλειά του. Τι άλλο να προσθέσω. Τα περισσότερα από αυτά που θα πω τα είπε και ο κύριος Κάσμαν. Ε, μια και μιλάμε για ποσοστά, υπάρχει και ο κίνδυνος ο όγκος της βοήθειας να μειωθεί τώρα με την κρίση. Επίσης, είναι περίεργο να φεύγουν τα λεφτά από τα συνήθη κανάλια και να τα βάζουμε στα αποθεματικά για να τα δίνουμε μέσα από ειδικά κανάλια. Δεν συμφωνώ πλήρως με αυτό λοιπόν. Επίσης, να προσθέσω κάτι άλλο. Για την κλιματική κρίση, που είναι τεράστια κρίση, χρειαζόμαστε επιπλέον κονδύλια γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν οι τάσεις στα κράτη-μέλη να λένε ούτως ή άλλως έχουμε την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια ε, για να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Πρέπει να τονίσουμε ότι δεν συμφωνούμε με αυτό. Για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναφέρθηκε και αυτό. Ούτως ή άλλως ε, τα περισσότερα δάνεια πηγαίνουν, επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μόνο το 0,6% πηγαίνει σε αφρικανικές χώρες. Αν θυμάστε την έκθεση της κυρίας Γουτζ του 2009, ε, ανέφερε ότι υπάρχει και το θέμα της αιρεσιμότητας, ένα διαρθωτικό πρόβλημα. Θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε στην έκθεση, ότι χρειαζόμαστε μια διαρθωτική μεταρρύθμιση, ούτως ώστε να είναι δυνατόν οι αναπτυσσόμενες χώρες να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια. Και επίσης ε, μην ξεχνάμε τις προτάσεις που έκαναν πρόσφατα ερευνητές που έλεγαν ότι το 1% του πακέτου κινήτρων στις αναπτυσσόμενες χώρες, στις αναπτυγμένες χώρες, συγγνώμη, θα μπορούσε να δοθεί στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ούτως ώστε να βοηθηθούν και αυτοί να αντιμετωπίσουν την οικονομική κρίση. Μήπως θα μπορούσε να μπει και αυτό στην έκθεση. Τα υπόλοιπα με βρίσκουν απόλυτα σύμφωνοι και σε ευχαριστώ για την έκθεση. Η Κομισιόν θέλει να απαντήσει. Ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ θα ήθελε να κλείσει παρακαλώ την ε, έκθεση. Πολύ σύντομα. Άκουσα τα ευνοϊκά σχόλια για την έκθεση, χαίρομαι γι' αυτό και θα ήθελα πολύ σύντομα να πω πρώτα το εξής. Καταρχάς, ότι η αρχική έμπνευση της έκθεσης αυτής ήταν η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο, που ήταν μια θαυμάσια έκθεση. Ε, χάρη σε αυτήν μπόρεσα και εγώ να εστιάσω ε, στα αναπτυξιακά θέματα. Ε, γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την έκθεσή της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας προειδοποίησε ότι η αντίδραση του Συμβουλίου δεν ήταν τόσο αρκετά ευνοϊκή όταν δημοσίευσε την έκθεσή της. Τώρα δεν θέλω να σχολιάσω με εμπριστικά σχόλια αυτή την έκθεση, δεν θέλω να είμαι εθνικιστής. Αλλά πιστεύω ότι επί Ισπανικής Προεδρίας στο Συμβούλιο, το Συμβούλιο θα είναι πιο ευνοϊκό για να προχωρήσει αυτή την πορεία δεν σας λέω ότι όλα όσα προτείνει η έκθεσή μου θα περάσουν, αλλά ως θέση και ως ε, διάθεση, ως φιλοδοξία κτλ. Τα έχουμε αυτά τα στοιχεία. Περιμένουμε την έκθεση της ε, Επιτροπής για τους ε, στόχους της χιλιετίας θα πρέπει να δουλέψουμε πολύ και επ' αυτής της ε, έκθεσης, ούτως ώστε πάλι κατά τη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας να αρχίζει να διαφαίνεται μια ευρωπαϊκή θέση ε, εν ώψη της ε, Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που το επόμενο φθινόπωρο θα αναθεωρήσει τους στόχους της χιλιετίας. Περιμένουμε με ανυπομονησία θα έλεγα λοιπόν αυτή την έκθεση. Τώρα, για αυτό που είπε ο κύριος ε, Κάσμαν. Δύο θέματα μπαίνουν εδώ. Το πρώτο, τα εμβάσματα για πολλές χώρες είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υπάρχουν χώρες όπου το 25% του ΑΕΠ τους προέρχεται από τα εμβάσματα. Είναι το τέταρτο έσοδο ετησίω των χωρών αυτών ή κάποιων χωρών. Επομένως είναι τεράστια σημασία. Κάτι άλλο που είπε και ο Μάικλ Κάσμαν και η κυρία Κέλλερ είναι το εξή. Ότι θα πρέπει, ή μάλλον είχα καταρχήν υπόψη μου να βάλω στην έκθεση ότι δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα ε, των ποσοστών όταν είμαστε σε φάση κρίσης. Γιατί η μείωση των, ε, του ΑΕΠ των αναπτυγμένων χωρών μπορεί να οδηγήσει στο εξή. Ότι αν κρατήσουμε απαράβλητο το ποσοστό της βοήθειας, τελικά θα δώσουμε λιγότερα κονδύλια στις χώρες αυτές. Επομένω πρέπει να τα δούμε τα πράγματα όχι με ποσοστά, αλλά με απόλυτε τιμέ. Ούτω ώστε σε απόλυτε τιμέ οι δεσμεύσει μα να μην μειωθούν. Τα, τα, ποσά συγγνώμη, που δίνουμε στην αναπτυξιακή βοήθεια να μην μειώνονται τελικά. Σε απόλυτε τιμέ, έτσι, όχι σε ποσοστά. Τέλο. Για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Είναι σαφέ ότι τα λεφτά που δίνουμε για να στηρίξουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες ε, να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν μπορούν να προέρχονται από τη σημερινή αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει να είναι νέοι πόροι. Πρέπει να είναι επιπρόσθετοι πόροι. Σε κάποια φάση είχα πει ότι στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του Σεπτεμβρίου ο Ισπανός Πρωθυπουργός πρότεινε να δημιουργηθεί ένα νέο ταμείο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής που θα εξυπηρετούσε στο να μεταφερθεί η τεχνολογία από εμά στις αναπτυσσόμενες χώρες για να ανταποκριθούν στις προκλήσεις και να καταπολεμήσουν τις κλιματικές αλλαγές. Οι απόψεις οι οποίες εκφράστηκαν θα αντικατοπτρίζονται και στην τελική εκδοχή του κειμένου. Αυτές οι απόψεις. Ευχαριστώ λοιπόν του συναδέλφους την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα λοιπά που υποστήριξαν σε γενικές γραμμές την έκθεσή μου και είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε. Will Ωραία. 1η Μαρτίου θα ψηφίσουμε για την έκθεση αυτή και 7 Φεβρουαρίου στις 6 το απόγευμα είναι η προθεσμία και κατάθεση τροπολογιών στην έκθεση αυτή που μόλις συζητήσαμε του κυρίου Γκερέρο Σαλόμ. Πάμε τώρα στο σημείο 10. Είναι η αντιπροσωπεία της Επιτροπής μας ως διευρετική αποστολή στο Μπαγκλαντές. Πριν από λίγες εβδομάδες πήγαμε. Εγώ ήμουν επικεφαλής της αντιπροσωπείας μας αυτής, πήγε στο Μπαγκλαντές. Και θα σας παρουσιάσω από εδώ, αν δεν έχετε αντίρρηση την ε, παρουσίασή μου. Εκτός αν θέλει κάποιος άλλος να έρθει εδώ να προεδρεύσει για να κατέβω εγώ να σας την πω από κάτω. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν στο Ντακάρ καταρχήν με τον πρόεδρο της αντιπροσωπείας ε, για την Νοτιοανατολική Ασία, Λάμπερτ, και με κάποια μέλη της ε, επιτροπής αυτής ε, και της αντιπροσωπείας της Νοτιοανατολικής Ασίας. Πήγαμε λοιπόν στο Μπαγκλαντές επειδή είναι μια από τις χώρες η οποία κεντρεύει περισσότερο από την αύξηση της στάθμης των υδάτων. Θέλαμε λοιπόν να δούμε πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά εκεί τις επιπτώσεις από τις αλλαγές στο κλίμα και να εκτιμήσουμε την κατάσταση αλλά και το τι έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Πέρα από τις κλιματικές αλλαγές και την αναπτυξιακή βοήθεια, συζητήσαμε και την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Υπήρξε και μία συνάντηση με τον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Συναντηθήκαμε με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου, τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον Υπουργό για την Διατροφή. Ε, συναντηθήκαμε επίσης με επικεφαλής της Αντιπολίτευσης και τους επικεφαλής των Αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκεί. Επίσης συναντηθήκαμε και με δωρητές, με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με οργανώσεις του ΟΗΕ. πήγαμε και 200 χιλιόμετρα πέρα από το Δάκα που είναι μια διαδρομή πολύ ενδιαφέρουσα θα έλεγα. Τα συμπεράσματά μας έχουν ως εξής. Επίγει να δράσουμε τώρα. Αν δεν αναλυθούν μέτρα άμεσα όσον αφορά τις προσαρμογές στις κλιματικές αραγές, με επιπλέον πόρους, με επιπλέον προγράμματα, τότε εκατομμύρια άνθρωποι θα αναγκαστούν να φύγουν από εκεί για να βρούν αλλού καταφύγιο, κάτι το οποίο θα δημιουργήσει βέβαια τεράστιες προκλήσεις στις ε, κοντινές εκεί χώρες, αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες. 30 εκατομμύρια περίπου άνθρωποι ξεκινούν να μετακινούνται. Θα υπάρξουν προβλήματα στην Ινδία, διαμάχες και Πολλοί έχουν συγγενεί στην Αγγλία για παράδειγμα. Πολλοί λοιπόν θα θελήσουν να έρθουν στην Ευρώπη από τους κατοίκους του Μπαγκλαντές. 20 εκατομμύρια άνθρωποι από ό,τι φαίνεται θέλουν να έρθουν στις χώρες μας. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να τους υποδεχτούμε. Πρέπει συνεπώς να δώσουμε στήριξη στον Παγκλαντέ. με επιπλέον χρηματοδότηση στα πλαίσια μάλιστα της διάσκεψη της Κοπεχάγης που λαμβάνει η χώρα αυτές τις μέρες. Η κυβέρνηση του Μπαγκλαντές προσπαθεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της αλλαγής του κλίματος με 100 εκατομμύρια δολάρια από το δικό της προπολογισμό για να προσαρμοστεί η χώρα με προγράμματα δράσης. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος έκανε έκκληση για άμεση χρηματοδότηση 10 δις αμερικανικά δολάρια προκειμένου να υπάρξουν προσαρμογές, προγράμματα, ώστε να ανυψωθούν ε, τα χωριά τα οποία κινδυνεύουν από το νερό, από πλημμύρες. Επίσης ε, θέλουν να αντλήσουν νερό από τα ποτάμια, να γίνουν κομματώσεις και φράγματα. Εμείς είδαμε τι χρηματοδοτείται, τι προγράμματα χρηματοδοτούνται, τα είδαμε τα προγράμματα αυτά επιτόπου, τι χρηματοδοτείται από εμά. Ένα χωριό, τρία εκτάρια, ανυψώθηκε, σηκώθηκε. 1,5 μέτρο κάτω από, μάλλον πάνω, βέβαια από το επίπεδο του νερού. Τρεις μήνες κράτησε το πρόγραμμα αυτό. Και το κάνανε οι ίδιοι οι κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι ανήψωσαν το επίπεδο του χωριού. Το σύνολο του κόστους για τα τρία αυτά εκτάρια ήταν 6.000 ευρώ. Πολλά χωριά λοιπόν πλημμυρίζουν συχνά και άρα το μισό χρόνο σχεδόν οι κάτοικοι δεν μπορούν να μείνουν εκεί γιατί είναι πλημμυρισμένα τα χωριά τους. Επιπλέον, πέρα από την ανύψωση αυτή, έχουν την γεωργική παραγωγή, έχουν κατσίκια, πρόβατα και άλλα, τα οποία προσπαθούν να τρέψουν για να μπορούν να βρουν τρόφιμα για τους αυτούς τους. Να λοιπόν ένα παράδειγμα τι μπορεί να γίνει για να υπάρξει αυτή η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Θα δώσω το λόγο βέβαια και σε συναδέλφους. Ε, όλοι εντυπωσιαστήκαμε κυρίως γιατί το κόστος ήταν πολύ χαμηλό. Βέβαια υπάρχουν 30.000 τέτοια χωριά στον Μπαγκλαντές που θα μπορούσαν να ανυψωθούν με τον ίδιο τρόπο, δύο μέτρα, για να μην πλημμυρίζουν. Αν τα τρία εκτάρια γίνονται για 6.000 ευρώ, ανυψώνονται, τότε με 100 εκατομμύρια ευρώ θα μπορούσαν να ανυψωθούν όλα τα χωριά που πλημμυρίζουν. Ο Πρωθυπουργός εκεί επίσης μας μίλησε για την εμβάθυνση των ε, ποταμών. ώστε να μην πλημμυρίζουν τα ποτάμια και πλημμυρίζουν και γύρω περιοχές. Αν βαθύνουν λοιπόν τα ποτάμια, θα υπάρχει περισσότερο περιθώριο για νερό. Όλα αυτά είναι πράγματα εφικτά. Είναι εξαιρετικά προγράμματα, σχετικά απλά, που συγκριτικά εύκολα μπορούν να τα κάνουν οι ίδιοι από μόνοι τους. Με λίγα χρήματα. Η κυβέρνηση επίσης ανησυχεί και για το θέμα ξαφνικών πλημμυρών που έχουμε, πριν από δύο χρόνια θυμάμαι εδώ, είχαμε συζητήσει με πρέσβεις από την Ινδία, την Κίνα, το Πακιστάν, Παγκλαντές, Νεπάλ. Ε, και από τον Πουτάν. Είναι σαφές ότι δεν μπόρεσε εκείνο μάλλον να έρθει τότε, τον είχαμε καλέσει αλλά δεν ήρθε. Είδαμε λοιπόν για το Γάγκη, το Κίτρινο Ποταμό, το Γεροποτή, το Τζάρα. υπάρχουν πάγοι οι οποίοι στέλνουν νερό στα ποτάμια αυτά, που επίσης λιώνουν σιγά σιγά. Είναι καταστροφική κατάσταση. 1,3 δις άνθρωποι ζουν στις περιοχές αυτές και θα έχουν όλο και λιγότερο νερό για να αρδεύουν τα, τους αγρούς τους. Οι παγετοί μειώνονται με ταχύτητα τρεις φορές παραπάνω από ό,τι έχουμε στον ε, Βόρειο και Νότιο Πόλο. Είναι ο τρίτος πόλος, έτσι λέμε αυτούς τους παγετούς, έτσι ονομάζονται. Και επηρεάζονται και αυτοί από παράγοντες που είναι καθαρά ανθρώπινοι. Γι' αυτό λοιπόν, συνάδελφοι, πρέπει να αναγνωρίσετε τη διάκριση που υπάρχει. Οι παγετοί δεν λιώνουν απλώς και μόνο εξαιτίας της θέρμανσης του πλανήτη, οι παγετοί αυτοί λιώνουν εξαιτίας του άνθρακα. Του λευκού άνθρακα όπως λέμε. Γιατί υπάρχει ο άνθρακας που έχουμε από το κάψιμο του ξύλου, ας πούμε για να θερμαθούν οι άνθρωποι στην Ιδία, στον Παγκλαντέ και αλλού, για να μαγειρέψουν. Και από εργοστάσια αηλεκτρισμού που πάει πάνω στους παγετώνες κατακάθεται και ο ήλιος πιο εύκολα επειδή δεν υπάρχει αντανάκλαση λιώνει τους παγετώνες αυτούς. Είναι διπλή λοιπόν η δράση, γι' αυτό και τα αποτελέσματα προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα. Αν θέλουμε να σταματήσουμε το πρόβλημα αυτό, πρέπει να σταματήσει και το λιώσουμε αυτών των παγετών. <clears throat> Όλος παραδόξως, αυτό το πρόβλημα που είπαμε ότι επηρεάζει 1,3 δισεκατομμύρια ανθρώπου στην Ασία, δεν υπάρχει στην ημερήσια διάταξη της Κοπεχάγης. Μιλάνε για εκπομπές, αλλά δεν μιλάνε για αυτό το πρόβλημα, το οποίο είναι μοναδικό φαινόμενο. Εμεί από τη δικιά μας την πλευρά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι μπορούμε να κάνουμε. Και έχουμε ηγετική θέση εδώ για να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές ε, και να μην συνεχιστεί το λιώσιμο των πακετών εκεί. Πολλοί στον Παγκλαντέ θέλουν να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους είναι πολύ πιο έτοιμοι να δράσουν από ότι άλλες, άλλες χώρες που έχω δει. Θέλουν να βοηθήσουν τους εαυτούς τους για να αποφύγουν αυτές τις καταστροφές που τους περιμένουν. Δεν λένε ελάτε να κάνετε εσείς τη δουλειά για μας, όχι θέλουν να την κάνουν οι ίδιοι. Αλλά χρειάζονται κάποια απλά μέσα, λίγα χρήματα για να αγοράσουν, να χρησιμοποιήσουν μέσα τα οποία θα τους βοηθήσουν να δουλέψουν και να προσαρμοστούν έτσι στις κλιματικές αλλαγές. Επίσης, νιώσαμε ότι χρειάζεται και συνεργασία στην περιοχή. Ιδίω για τα Ιμαλάγια, τους πακετώνες δηλαδή των Ιμαλαίων. Οι Κινέζοι και οι Ινδοί, οι Κινέζοι για παράδειγμα, σκοπεύουν να φτιάξουν φράγματα ε, σε ένα ποτάμι στο Θηβετιανό πλατό. Κάτι το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό για τις πλημμύρες που έχουν συχνά. Αλλά πρέπει να προσέξουν να μην υπάρξει σύγκρουση εκεί. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι την περιοχή αυτή την έχουμε αγνοήσει εμείς, την έχουμε αφήσει στην τύχη της, όχι επίτηδες, αλλά γιατί ασχολούμαστε πάρα πολύ με τις χώρες, ΑΚΕ δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες, αλλά πάρα πολλοί κόσμος ζει εκεί στην Ασία και πρέπει να δράσουμε τώρα. Και το εννοώ. Πρέπει να δράσουμε τώρα. Πριν υποστούμε μεταναστευτική πίεση και πρόσφυγες από εκεί. Θέλω να ολοκληρώσω γιατί βέβαια έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε. Αλλά θέλω να δώσω το λόγο στους συναδέρφους που ήταν μαζί για να σχολιάσουν ή τους υπόλοιπους για να σχολιάσουν το όσα εγώ είπα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, ευχαριστώ τον Πρόεδρο Δέδε για το πώς ηγήθηκε αυτή της αντιπροσωπείας με έναν τρόπο τρομερά αποτελεσματικό. Η αντιπροσωπεία μας λειτουργήσε με συνενετικό τρόπο καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης στο Μπαγκλαντές. Συμφωνώ με την ανάλυση που έκανε <clears throat> ενώπιον των μελών της Επιτροπής. Θέλω να προσθέσω τέσσερα στοιχεία τα οποία εντάσσονται στα όσα είπε ο πρόεδρος Δέβα. Το πρώτο, θα ήθελα να σας δώσω κάποια αριθμητικά στοιχεία από αυτή τη χώρα. Ο κύριος Δέβα ανέφερε κάποια αριθμητικά στοιχεία. Είναι μια χώρα όπου 20 εκατομμύρια ανθρώπων μπορεί να ζητήσουν όχι πολιτικό άσυλο, αλλά κλιματικό άσυλο σε αυτή την, στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια, την επόμενη ε, δεκαετία είναι ένα τεράστιο νούμερο που μας το δίνουν ε, βρετανικές πηγές. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε. Μιλάμε για μια χώρα όπου το 20% της έκτασής του κινδυνεύει να βυθιστεί στο νερό σε περίπτωση που υπάρξει αύξηση της στάθμης. Ε, κατά 0,8 μέτρα των νερών της θάλασσας. Μια χώρα όπου το 50% του πληθυσμού είναι κάτω των 15 ετών. Μια χώρα όπου το 30% των 150 εκατομμύριων κατοίκων δεν έχει τις απαραίτητες θερμίδες. Δηλαδή υποσυτίζεται καθημερινά. Νομίζω ότι αυτά τα νούμερα και τα συζητήσαμε με τους εκπροσώπους της Επιτροπής και τους πρέσβης, θα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο μιας στρατηγικής επικοινωνίας για να μιλήσουμε για αυτό το πρόβλημα, για να δημιουργήσουμε μια ε, συνείδηση του τι σημαίνει η τι αντιμετωπίζει το, το τι προβλήματα, τι κινδύνου. Αυτά τα νούμερα θα πρέπει να γνωστοποιηθούν, θα πρέπει να τα ψάξουμε, θα πρέπει να τα διαδώσουμε στον κόσμο έτσι με τρόπο στρατηγικό, ούτω ώστε να τα καταλάβουν, να τα καταλάβει το κοινό. Δεύτερο, όπως είπε και ο κύριος Ντέβα, είναι μια χώρα όπου ε, φύγαμε με κάποιες ελπίδες. Γιατί υπάρχουν μια σειρά από προγράμματα ε, μικροπρογράμματα θα έλεγα, ευαισθητοποίησης του πληθυσμού, του τοπικού πληθυσμού. Ε, υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες έτσι, αυτοπροστασίας των πολιτών. Οι κάτοικοι μαθαίνουν να δρουν. Και με αυτόν τον τρόπο μειώθηκαν δραστικά ε, τα θύματα του τελευταίου κυκλώνα. Αυτό ήταν πολύ ελπιδοφόρο. Τρίτον, θα να μην ξεχνάμε ότι το Μπαγκλαντές είναι μια χώρα πολύ μεγάλη, από τις πιο μεγάλες ε, σε μουσουλμανικό πληθυσμό. Είναι η τρίτη μουσουλμανική χώρα στον πλανήτη. Και είναι μια χώρα όπου αντιμετωπίζει κάποια στερεότυπα και επιβεβαιώνει τα στερεότυπα που υπάρχουν ε, στους Ευρωπαίους. Ότι το Ισλάμ είναι ασυμβίβαστο με μια λειτουργούσα δημοκρατία, ε, το Ισλάμ είναι ασυμβίβαστο με τις γυναίκες ε, ενεργές και δραστήριες. Έχουμε μια κουτσή δημοκρατία στο Μπαγκλαντές. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια δημοκρατία. Αυτή η κουτσή δημοκρατία και που επιτρέπει μια εναλλαγή στην εξουσία. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να προκύψει ένας πραγματικός πολιτικός πλουραλισμός. Ε, επίσης, ο Πρωθυπουργό είναι ε, γυναίκα. Αλλά και έχουμε και πολλούς υπουργού γυναίκες. Και πολλές γυναίκες υπάρχουν και στην αντιπολίτευση. Επομένως, Όλα αυτά θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και να τα προωθήσουμε για, και να καταλάβουμε ότι η χώρα αυτή δεν αποτελεί μόνο στερεότυπα, αλλά έχει ξεπεράσει και κάποια στερεότυπα. Ένα τέταρτο σημείο, το οποίο δεν ανέφερε ο πρόεδρος Ντέβα και το οποίο το συζητήσαμε όταν ήμασταν στον Μπαγκλαντές, είναι το εξής. Τα νούμερα λένε ότι σε λίγο το 50% του πληθυσμού θα ζει σε αστικές περιοχές. Εγώ έζησα δύο χρόνια στην Ασία, σε εκείνη την περιοχή, μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν. Αλλά το να κινείται κανείς στα δρομάκια της Ντάκα είναι απίστευτο. Ε, είναι ένα χάος έτσι, αστικό. Υπάρχει απίστευτος πληθυσμός, ε, απίστευτος κόσμος. Ε, σχεδόν σε πνίγει αυτός ο πληθυσμός με μια άτυπη οικονομία, έτσι, αστική, που δεν αναγνωρίζεται, που δεν είναι νόμιμη, αλλά που υπάρχει στα, ενώπιον όλων. Ε, περίπου το 70% της οικονομικής δραστηριότητας της πόλης και επομένως τελικά και της χώρας γίνεται χωρίς καθόλου ε, υπηρεσίες, χωρίς αποχέτευση, χωρίς ε, αστικό σχεδιασμό, χωρίς ε, ιατρία σε διάφορες γειτονιές και αυτό είναι το πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει μια φοβερή έτσι, αδιαφορία από πλευρά διεθνού κοινότητα. Εμεί επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ στην ανάπτυξη των αστικών περιοχών, ε, μιλάμε για κοινωνικές υπηρεσίες ε, της αλλά σε αυτή τη χώρα, όπως ε, μετά από τις συζητήσεις που είχαμε με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τους πρέσβεις, με την Κομισιόν κτλ, δεν υπάρχει μια δράση α, συνεργασίας στον αστικό ιστό. Αυτό ισχύει όχι μόνο για τον Μπαγκλαντές, αλλά και για άλλες χώρες. Η, χώρα αυτή ε, ζει ανάμεσα στις δύο μεγαλοπόλεις, την Τάκα και την Τόκ. Θα πρέπει το πούμε αυτό το γεγονός. Θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν να παρέμβουν με δράσεις στοχευμένες, με μικροπιστώσεις, για να αναπτυχθούν ε, διάφορες γειτονιές, με μικρές υποδομές που βοηθάνε τις αστικές περιοχές. Δεν θα πρέπει επίσης μόνο να ασχοληθούμε με τις αποχετεύσεις στην ΤΑΚΑ, αλλά γενικά με όλα τα ζητήματα υγιεινής. Ε, αυτό που λέμε στα αγγλικά water and sanitation, δηλαδή νερό και αποχετεύσεις. Ευχαριστώ. Μου άρεσε πραγματικά, Νίκολα, ε, το ταξίδι μας και όλα αυτά ήθελα να τα διαμηνήσω στους συναδέλφους. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης, γιατί θα έρθει σε λίγο ο προσκεκλημένος μας και πριν έρθει θα ήθελα ο κύριος Κάσμαν, που είναι ο, ο υπεύθυνο για την επόμενη έκθεση, να μας μιλήσει, γιατί μετά έχουμε τον Πρωθυπουργό του, του, Βαλιού, του Βαλού. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μια σύντομη προφορική έκθεση. Γραπτή έκθεση θα καταθέσω τον Ιανουάριο στην Επιτροπή. Με χαρά βλέπουμε από την αντιπροσωπεία αλλά και την ημερήσια διατάξη τη δέσμευση για ε, περισσότερη σκληρή δουλειά που βλέπετε και εσείς γιατί πολλές φορές αυτές οι αντιπροσωπείες χαρακτηρίζονται από τον τύπο ως μια ευκαιρία για ε, ευχάριστες διακοπές σε κάποιο συμπαθητικό θέρετρο για τους ευρωβουλευτές. Οι συνάδελφοι θα σας βεβαιώσουν για το αντίθετο, ότι έχει πολύ σκληρή δουλειά μια τέτοια αποστολή. Θα ήθελα να ευχαριστώ την κυρία Νίκα Βασιλεύα και την κυρία Νίκα Λουόμα που μας συνόδευσαν από την γραμματεία και, ε, και σκληρά εργάστηκαν και πριν να ξεκινήσουμε εμείς τη δουλειά μας και αφότου εμείς είχαμε τελειώσει. Τις ευχαριστούμε λοιπόν. Ο κύριος Φίλιπ Καζαμάρεκ και ο υποφαινόμενος, ως επικεφαλής, ο κύριος Αργεντίνη, η κυρία Θεοχάρους που είναι και εδώ μαζί μας ήταν μέλη της αντιπροσωπείας. Τους ευχαριστώ για τη σκληρή δουλειά και την αντιπροσωπεία. Είχαμε ίσως, ε, έχουν κάποιοι συνάδελφοι ανάμνηση από τον εκπρόσωπο που συναντήσαμε εκεί πέρα, από συνεδριάσεις που ερχόταν στο παρελθόν, ήταν παρόν λοιπόν και με το προσωπικό του, ο της Επιτροπής μας ενημέρωσε ε, και ήταν στη θέση μας για κάθε πρόβλημα. Ο κύριος Μαρκ Τίλ ήταν παρόν επίσης για την συνολική ενημέρωση, όπως και εκπρόσωποι από τις πρεσβείες των, των ευρωπαϊκών κρατών, ο εκπρόσωπος ε, ε, από το Ηνωμένο Βασίλειο, εκπρόσωπος από την Γαλλική Πρεσβεία, ο πρέσβης της, των Πολιτειών και της Γερμανίας, εκπρόσωποι της Παγκόσμιας Τράπεζας του, του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών. Όλους ε, αυτούς θα τους δείτε και στο προσάρτημα στο κείμενο όταν δείτε την γραπτή έκθεση. Ξεκινήσαμε με επαφές με την ε, κοινωνία των πολιτών μαζί και με την οργάνωση Μποκόγκο που είναι η Ομοσπονδία θα έλεγα ε, συστήσαμε θέματα από τα δικαιώματα των γυναικών, την ισότητα των φίλων, ε, τα παιδιά, την νεολαία, την, την εκπαίδευση, πρόσβαση στην εκπαίδευση. Είδαμε εκπροσώπους του εμποροβιομηχανικού κλάδου αλλά και των ενώσεων των βιοτεχνών. Από την κυβέρνηση είδαμε τον Αντιπρόεδρο Μιουφάγη τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, την πρόεδρο Μάργκριτ Νάσσερ και μάλιστα σας συνιστώ να παρακολουθήσετε πώς είναι σε θέση να ελέγχει μια ομάδα βουλευτών η κυρία Νάσσερ σε μια συνεδρίαση, τα καταφέρνει εξαίρετα με σιδηρά πυγμή και βέβαια είναι η πρώτη γυναίκα πρόεδρος κοινοβουλίου στην Ποτσουάνα. Είδαμε επίσης τον Υπουργό Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Βιομηχανίας, Εξωτερικών, τον εκτελεστικό γραμματέα της ΣΑΝΤΑΚ, με πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση ως προς τις ε, ενδιάμεσες συμφωνίες και τη δυνατότητα για ευρωπαϊκή, ε, είτε ο, ε, κατά το ευρωπαϊκό σύστημα περιφερειακή ολοκλήρωση ή, ή αντίθετα περιφερειακή αποδιάρθρωση. Ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα ήταν ότι οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις είναι ιδιαίτερα ενήμερες για τις ενδιάμεσες οικονομικές συμφωνίες σχέσεις, Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για αυτές. Ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για, τις, ε, για την οδηγία περί υπηρεσιών. Τους διαβεβαίωσα γιατί ότι αυτή η οδηγία εξασφαλίζει και πρόσβαση στις, οδηγίες, στις ε, υπηρεσίες για υπηκόους ξένων κρατών. Μιλήσαμε δηλαδή πολύ για την οδηγία Bolkenstein, επίσης μιλήσαμε πολύ για την ρήτρα και το καθεστώς του ε, μάλλον ευνοούμενου κράτους και ιδίω για αυτή την, ε, οικονομική, εταιρική οικονομική σχέση είδαμε ότι η Μποτσουάνα ενδιαφέρεται περισσότερο, άλλωστε αυτό είδαμε από, τις, από όλους τους συνομιλητές μας στην Μποτσουάνα, για μια ολοκληρωμένη πλήρη ΕΠΑ και όχι μόνο για μια προσωρινή. Ναι. Πολύ χρήσιμη λοιπόν αυτή η συνάντηση. Επίσης είδαμε και τον ε, επικεφαλής της Εθνικής ε, Οργάνωσης του Εθνικού Φορέα Τονισμού για το AIDS με τις προσπάθειες για την εξασφάλιση υπαρκών ποσοτήτων φαρμάκων ε, κατά του ιού για τους φορείς και εν γέννη θα έλεγα ότι γιατί δεν έχουμε χρόνο ήταν πολύ παραγωγική η επίσκεψη κράτος το οποίο θεωρείται ότι είναι μέσου εισοδήματος. Είναι χρήσιμο να δούμε πώς αντιμετωπίζει την οικονομική κρίση. Η Μποτσουάνα έχει κυρίως διαμάντια, άνθρακα και χαλκό. Νικέλιο, συγγνώμη, και χαλκό ως εξαγωγικά προϊόντα. Και τώρα με τις γιορτές που έρχονται τα Χριστούγεννα την Πρωτοχρονιά, του Αγίου Βαλεντίνου, το την Κινέζικη Πρωτοχρονιά που αποτελούν για μας σταθμού στη ζωή μας, ε, εκείνοι περιμένουν να δουν τις ενδείξεις περί διαφυγής από την κρίση, δηλαδή τα, τα χρονικά σημεία στο δικό μας ημερολόγιο στα οποία κάνουμε τις ε, πολυτελείς μας ε, αγορές ή δαπάνες, για αυτούς είναι σημεία καμπή. Και πρέπει να σας πω ότι η πόλη των διαμαντιών είναι για αυτούς πολύ ε, χρήσιμη επιχείρηση. Έχουν καταφέρει να αναπτύξουν τεράστια οικονομικά αποθέματα χάρη στην πώληση των διαμαντών και ταυτόχρονα προστατεύουν και τις επενδύσεις τους ε, σε ε, ομόλογα κτλ ένα μέρος του προπολογισμού του το 1 τρίτο, πηγαίνει στην εκπαίδευση. Χώρα η οποία τόσο πολύ εξαρτάται από τον Νικέλιο, το Χαλκό και τον Αδάμαντα, ε, ενδιαφέρεται και στρέφεται ιδιαίτερα προς την ε, διαφοροποίηση ξέρει ότι χωρίς σωστή εκπαίδευση και διαφοροποιημένες δεξιότητες δεν θα μπορέσει να αναπτύξει την οικοδομία της και ταυτόχρονα τον προϋπολογισμό της και για το AIDS, HIV, τα φάρμακα που χρειάζονται και για την πρόληψη του τον, τον χρησιμοποιεί και ενδιαφέρον είναι ότι όσοι χρειάζονται αυτά τα αντικαφάρμακα, φάρμακα κατά 85% εξασφαλίζουν τα φάρμακα κατά το ιού του AIDS. 85%. Σε αξία εμπορική αγοράζω τα φάρμακα στην ε, αγοραία τους αξία. Και ενώ υπάρχει ένα έλλειμμα 4% στον προϋπολογισμό, μπορούν να δανειστούν λόγω της, των αξιό, της αξιοπιστίας τους, της δανειοληπτικής τους πίστης ε, που στηρίζουν στα τεράστια αποθεματικά τους. Αλλά όπω είπαμε και νωρίτερα, τα αποθέματα μερικέ φορέ καλό είναι να αξιοποιούνται, να απορροφούνται και θα πρέπει αυτό το θέμα να το παρακολουθήσουμε. Ήταν ιδιαίτερα λοιπόν χρήσιμη και ε, θετική αυτή η εμπειρία. Ήταν μια πηγή αισιοδοξία στο να δω ότι υπάρχουν άνθρωποι, πολιτικοί, κυβερνήτε, ε, ηγέτες οι οποίοι ασχολούνται με τη χώρα του, με το λαό του, θέλουν να αντιμετωπίσουν τι μεταναστευτικέ ροέ από χώρε όπω η Ζιμπάμπουε κατά τρόπον ανθρωπιστικό σε κάθε επίπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν ότι χωρίς εκπαίδευση δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Υπάρχουν άνθρωποι που βλέπουν ότι η γυναίκα και η πρόσδοση ικανοτήτων χειραφέτης της γυναίκας θα μπορέσει να δώσει μια πιο ισότιμη κοινωνία. Αισθάνομαι ιδιαίτερη περηφάνεια για τη δουλειά που έχουν κάνει στην Ποτσουάνα και ιδιαίτερα με ανησυχεί το πρόβλημα της, ε, του λοιμού εντό αγωγικών χορηγών, της απουσίας δηλαδή χορηγών, ιδιαίτερα για χώρες ε, όπως η Ποτσουάνα που διαθέτει πόρους για να στηρίξει άλλες χώρες. Πολλές ευχαριστήσεις λοιπόν που έχω να εκφράσω και προς τους ε, ε, Μποτσουανούς που συνάντησα και προς τα μέλη της αντιπροσωπείας που με τίμησαν με την παρουσία τους και τη συντροφιά τους τη γραμματεία, η Ελένη ίσως να θέλει να πει και εκείνη δύο λόγια. Ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι ήταν τόσο πολλοί οι δημοσιογράφοι που εμφανίστηκαν στην ε, συνέντευξη τύπου και πόσο ενήμεροι ήταν και για τη δουλειά μας και για, τα, για τις ε, οικονομικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης και για τις για τον αντίκτυπό τους στις χώρες της περιοχής. Αυτά είχα να πω και πρόεδρε, όπως και εσείς, αισθάνθηκα ιδιαίτερη τιμή που ήμουν επικεφαλής αυτής της και διδάχθηκα πολλά από την επισκεψή μου. Ευχαριστώ και πριν ζητήσω από την κυρία Θεοχάρου να λάβει το λόγο, λέει ο κύριος Δέβα, εντυπωσιάζομαι με τόσα, από τόσο είπες, Μάικλ. Έκθεση υποδειγματική για μια χώρα υποδειγματική. Γιατί λοιπόν να μην έχουμε κοινέ εμπειρίε. Γιατί να μην μοιραστούμε αυτέ τι εμπειρίε με άλλε χώρε και να έχουμε κοινέ ε, και να βοηθήσουμε και του άλλου να δαχθούν από την εμπειρία και από τι προσπάθειε τη Μποτσουάνα. Με το ζήτημα των πρακτικών. Κύριε Θεοχάρου, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θέλω να τονίσω ότι ήταν μια εξαιρετική αποστολή και αυτό οφειλόταν βεβαίως τόσο στην κρατική υποδομή που υπάρχει στην ε, Μποτσουάνα, αλλά και στην εμπνευσμένη ηγεσία της αποστολής από τον Μάικολ Κάσμαν. Καλύψαμε σχεδόν όλους τους τομείς της αναπτυξιακής, ε, όλους τους αναπτυξιακούς τομείς στη χώρα αυτή όσον αφορά το κράτος, την οικονομία, την κοινωνία Βεβαίως κάποια από τα στοιχεία που μας εδόθησαν και τα ανέφερε πριν από λίγο ο Μάικολ χρήζουν κάποιας ανάλυσης και επιβεβαίωσης όπως για παράδειγμα η συμπεριφορά του κράτους απέναντι στους Μπούσμεν, το, η έννοια της εσωτερικής μετανάστευσης, της υποχρεωτικής μετανάστευσης από τις γύρω χώρες, της εκπαίδευσης, της υγείας και ε, κάποια άλλα. Ε, ο... ήθελα να σταθώ στο γεγονός ότι ο Μάικολ Κάσμαν ήταν ιδιαίτερα μετριοπαθής στην παρουσίαση του τρόπου με τον οποίο ηγήθηκε αυτής της αποστολή, Εμένα να μου επιτρέψετε να σας πω ότι διεύθυνε με εξαιρετική επιτυχία όλες τις συζητήσεις, μη επιτρέποντας να εκτρέπεται η συζήτηση προς άλλες κατευθύνσεις και ο κάθε, το κάθε μέλος είχε τη δυνατότητα να εκφράσει την άποψή του και να δώσει την δική του εκδοχή. Θα ήθελα ακόμα να σταθώ στο γεγονός ότι με το ίδιο πάθος που υπερασπίστηκε σήμερα το πρωί τα ανθρώπινα δικαιώματα και επέμενε ότι δεν μπορούμε να έχουμε τάπολ or multiple standards στην εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κανένα μέρος του κόσμου ούτε για τις αναπτυσσόμενες, ούτε για τις αναπτυγμένες χώρες, ούτε για αυτές που είναι σε ενταξιακή πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε για αυτές τις οποίες προσφέρουμε αναπτυξιακή βοήθεια ως Ευρωπαϊκή Ένωση, με το ίδιο πάθος υπερασπιζόταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και στην Ποτσουάνα. Και το λέω αυτό και επιμένω, γιατί κάποιοι από τους συναδέλφους μας, χτες συγκεκριμένα, στη συζήτηση με την Μικτή Επιτροπή της Τουρκίας, μας είπαν, και επίτρεψε μου Μάικολ να το πω αυτό, Μα είπαν «Ευαρεθήκαμε να σα ακούμε εσά να μιλάτε για τον Κυπριακό και για την Κύπρο». Αυτό σημαίνει double standards όσον αφορά την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αν κάποιοι συνάδελφοι ευαρέθηκαν, εμεί ευαρεθήκαμε να ζούμε αυτή την τραγωδία και αυτή την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για αυτό που είσαι και για τον αγώνα που κάνεις. Εάν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή σχόλια, θα μας πει ο κύριος Κάσιμαν, θα καλωσορίσω τον Πρωθυπουργό του Τουβαλού, Αγαπητοί συνάδελφοι, μεγάλη τιμή και χαρά για μένα. Το ότι είμαι σε θέση να καλωσορίσω τον κύριο Τσίμαγια, πρωθυπουργό του Τουβαλού, για να συζητήσουμε την ε, κλιματική αλλαγή. Ήδη συζητήσαμε ε, νωρίτερα την ε, κλιματική αλλαγή και τις πτυχές της που αφορούν τις Μαλδίβες και το Βαγκλαντές. Η συζήτηση με τον κύριο Πισάη Ελέμια βέβαια έρχεται στην κατάλληλη στιγμή καθώς ε, διεξάγονται ταυτόχρονα και οι, κλιματικές, ε, οι συζητήσεις για τις κλιματικές, κλιματικές αλλαγές στην Κοπενχάγη από τις οποίες περιμένει ολόκληρος ο κόσμος θετική έκβαση και κυρίως χώρες όπως το Τουβαλού που πλήγονται ιδιαίτερα από τις κλιματικές αλλαγές. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει πολλέ ε, μελέτες από τους ειδικού και του επιστήμονες στο παρελθόν. Μπορεί το τοβαλού να μην προσφέρεται για αντιπαραθέσεις επιστημονικές, αλλά πάντω είναι στην πρώτη γραμμή του κινδύνου ω προ την κλιματική αλλαγή. Και αν αλλάξουν οι κλιματικές συνθήκες και αυξηθεί το επίπεδο της θάλασσας, το τουβαλού κινδυνεύει ακόμη και από εξαφάνιση. Και ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Κύριε Πρωθυπουργέ, Κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στην Επιτροπή μας και που θα μας απευθύνετε το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί βουλευτές, αγαπητά μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τα θερμά σας λόγια και ευχαριστώ όλα τα μέλη της Επιτροπής για την ευκαιρία που μου δίνετε να ανταλλάξουμε απόψεις μέσω της σημερινής συνάντησης. Το Τουβαλού και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ε, θερμές ε, σχέσεις, μια εταιρική σχέση εδώ και πολλά χρόνια και η κυβέρνησή μου δεσμεύεται να εμβαθύνει και να ενδυναμώσει αυτή τη σχέση τα επόμενα χρόνια. Ένα από τα μεγάλα θέματα που επηρεάζουν την χώρα μας και απειλεί ούτως ή άλλως την ανθρωπότητα στο μέλλον είναι η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και οι κλιματικές αλλαγές. Σήμερα ήθελα να σας πω ότι ανησυχεί η χώρα μου για αυτό το παγκόσμιο πρόβλημα. Το Τουβαλού είναι, ε, ανήκει σε ένα τμήμα νησιωτικών εθνών που έχουν χαμηλή στάθμη και που θα αντιμετωπίσει πρόβλημα εάν αυξηθεί η στάθμη των υδάτων. Ε, αυτό απειλεί την ύπαρξη του έθνους μας. Όταν υπάρχουν ε, παλήριες, το θαλάσσιο νερό θα μπορούσε να φτάσει βαθιά μέσα στην, ε, στη γη μας και σε πολλές περιοχές καταστρέφει δέντρα και καλλιέργειες. Το θαλάσσιο νερό επίσης μπαίνει στον υδροφόρο ορίζοντα και φυσικά όπως σας είπα καταστρέφει καλλιέργειες και δέντρα. Η αύξηση της στάθμης και οι καταιγίδε ε, μειώνουν ε, τους περιορισμένους πόρους μας, τα δέντρα μας προστατεύουν από τις ε, καταιγίδε. Τα κοράλια μας πεθαίνουν εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας των υδάτων και επηρεάζουν το ευπαθές αυτό οικοσύστημα και την παροχή νερού ε, μη αλμύρου νερού. Έχουμε ε, όλο και μακρότερες, ε, μακρότερες περιόδους εξηρασίας, κάτι που μας δημιουργεί πρόβλημα σε ό,τι αφορά το νερό. Για να αποφύγουμε τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών θα πρέπει να αναλάβουμε δράση πάρα αυτά, ούτως ώστε να μειωθούν οι εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο. Όλες οι χώρες, νομίζω, θα πρέπει να κάνουν συγκεκριμένες προσπάθειες σε όλες τις υπήρους για να μειώσουν τις εκπομπές τους. Όλες οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να προωθήσουν διάφορα πακέτα ούτω ώστε μέχρι το 2017 να μειώσουν τις εκπομπές τους. Οι μεγάλες οικονομίες ε, θα πρέπει να προωθήσουν ε, πακέτα πέρα από τη, συνηθισμένη επιχειρηματική δραστηριότητα και οι αναπτυσσόμενες χώρες επίσης εθελοντικά θα πρέπει να λάβουν δράσεις για να μειώσουν τις εκπομπές τους. Για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου σε επίπεδα αποδεκτά, θα πρέπει να φτάσουμε το ανώτατο όριο των εκπομπών το 2015 και να υπάρξει μείωση μετά. Μετά θα πρέπει να μειωθούν δραματικά μετά το 2015. Μια παγκόσμια προσπάθεια για να μειωθούν οι εκπομπέ θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι η αύξηση θερμοκρασία του πλανήτη φτάνει το πολύ στο 1,5, ε, στο 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με, τα, με τις θερμοκρασίες που υπήρχαν πριν τη βιομηχανική εποχή. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες και αυτές περιλαμβάνουν καταρχάς την προσαρμογή και την ανάπτυξη φυσικών αμυνών, εθνικά προγράμματα προσαρμογής, τα λεγόμενα ΝΑΠΑ, τα οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν στα βασικά του στοιχεία. Η πρώτη προτεραιότητα είναι να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο άμυνας ε, στο Τουβαλού για να προστατεύσουμε την ακτογραμμή μας και τα, κοράλ, και την, ε, και τα κοράλια μας. Επίσης, ε, από εδώ και πέρα θα αντιμετωπίζουμε πιο σοβαρούς κυκλώνες. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε την κατάλληλη υποδομή για να προστατεύσουμε τον πληθυσμό, την περιουσία μας και τα ζώα μας από τις επιπτώσεις των κυκλώνων. Επίσης, τρίτον, δεσμευόμαστε να μειώσουμε τις δικές μας εκπομπές, παρότι είναι απειροελάχιστη σε σχέση με αυτές άλλων χωρών. Έχουμε προωθήσει ένα πακέτο με την χρήση ανεώσιμων πηγών ενέργειας ε, μέχρι το 2020. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι Ευρωπαίοι ηγέτες έχουν πάρει το προβάδισμα σε αυτή τη μάχη για να βοηθήσουν τις πιο ευπαθείς χώρες. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα μέλη του Κοινοβουλίου και τον κύριο Τάνο Κόλος Ιδιωτέρος για το προφορικό ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση προς τα αναπτυσσόμενα μικρά νησιωτικά κράτη ε, μέσω του ΣΥΤΕΣ. Η απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ διαφωτιστική. Ε, με βάση τη συμμαχία ε, που δημιουργείται για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών, τα 3,2 εκατομμύρια θα πάνε στο Βανουάτου και στις ε, Μαλδίβες, στα πλαίσια πιλωτικών προγραμμάτων. Επίσης, οι Μαλδίβες παίρνουν 2,2 εκατομμύρια ευρώ για την περιφερειακή ανάπτυξη, για να προωθήσουν ένα τρόπο ζωής ε, πιο φιλοπεριβαλλοντικό. Επίσης, ε, στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας, ε, τα χρήματα δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούν μη βιώσιμα προγράμματα. Εμείς αντιμετωπίζουμε ένα αβέβαιο μέλλον λόγω των κλιματικών αλλαγών. Εμείς θα θέλαμε να παραμείνουμε εκεί που είμαστε, να συνεχίσουμε να υπάρχουμε, να διατηρήσουμε τον τρόπο ζωής μας, τον πολιτισμό μας. Δεν σκοπεύουμε να φύγουμε από το τουβαλού. Αν ληφθούν οι κατάλληλες δράσεις για να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές, θα παραμείνει ζωντανό το τουβαλού. Αν η Κομισιόν φοβάται ότι η βοήθεια προς, την, προς το τουβαλού μπορεί να μην είναι βιώσιμη, ε, νομίζω ότι θα έπρεπε να λάβει υπόψη της το ε, καταπίστευμα που έχουμε δημιουργήσει ε, για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των κλιματικών αλλαγών. διάφοροι δωρητές έχουν δώσει κονδύλια σε αυτό το, έχουν συνεισφέρει σε αυτό το καταπίστευμα. Ε, μας βοηθάει επίσης ε, σε επίπεδο προϋπολογισμού το Ηνωμένο Βασίλειο και επίσης μας βοηθάει ε, για διάφορα προγράμματα όπου δεν υπήρχαν καθόλου δωρητές. Με βάση την Διεθνή Συμφωνία για το Καταπίστευμα, κάθε δεκάρα που συνεισφέρουν οι δωρητές ελέγχεται από αυτούς. και τα χρήματα, η συνεχεία, πραγματικά πηγαίνουν στο τουβαλού. Το καταπίστευμα αυτό δημιουργήθηκε το 87 με 10,6 εκατομμύρια δολάρια. Αυστραλέζικα δολάρια. Τώρα έχουμε ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια. Με χρόνο και υπομονή το αυξανόμενο εισόδημα από το καταπίστευμα θα μπορούσε ε, να χρηματοδοτήσει διάφορα προγράμματα τα οποία δεν θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν οι δωρητές για να αντιμετωπίσουμε την ε, κλιματική αλλαγή. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με αφήσατε να μιλήσω για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε λόγω κλιματικής αλλαγής και με μεγάλη χαρά θα απαντήσω σε οποιαδήποτε ερωτήματα έχετε. Ευχαριστώ και εγώ σε ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ για την ε, ειλικρινή σας δήλωση. Είμαι ευρωβουλευτής εδώ και πολύ καιρό. Αλλά δεν είχα ακούσει αυτά που είπε ο Επίτροπος για το μέλλον της χώρας σας. Νομίζω ότι δεν ήταν σωστά αυτά που είπε ο Επίτροπος. Και πριν μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Κάσμαν. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ. Που ήρθατε να μας μιλήσετε για την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειες της. Κάποιοι ίσως να λένε ότι δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή. Ή κάποιοι μπορεί να λένε ότι οι ανθρώπινες δραστηριότητε δεν την έχουν προκαλέσει. Όμω εσεί μα υπενθυμίζετε με την παρουσία σα εδώ ότι είναι πολύ διαφορετική και σκληρή η πραγματικότητα. Εδώ πολύ συχνά συζητούμε τι επιπτώσει τη κλιματική αλλαγή σε μικρέ νησιωτικέ χώρε. Ε, μερικές, αυτό όμως μας απασχολεί όμως συνήθως μόνο στις ε, στιγμές της κρίσης, ε, την ώρα που βλέπουμε τραγικές επιπτώσεις. Εσείς όμως με την παρουσία σας εδώ μας υπενθυμίζετε ότι είναι σωρευτικό το φαινόμενο, ότι είναι διαρκές το φαινόμενο και ότι έχει πολλές ε, πτυχές και διαφορετικούς τρόπους εκδήλωσης, γιατί έχει και πολύ έντονες βροχοπτώσεις και πολύ έντονες ξηρασίες και κινδυνοποίθησης ή ανόδου της ακτογραμμής. Όλοι συμφωνούμε ότι χρειάζεται συμφωνία στην Κοπενχάγη, όλοι ε, συμφωνούμε ότι χρειάζεται δέσμευση όχι μόνο στα λόγια, αλλά και με κονδύλια τα οποία θα υλοποιηθούν για την εκτέλεση των δεσμεύσεων της Κοπενχάγης. Ναι, θα πρέπει να εξασφαλιστεί ο περιορισμός των, ε, των εκπομπών το 2017, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει μέχρι το 2015 να αφήσουμε ανεξέλεκτες ε, τις εκπομπές. Κύριε Πρωθυπουργέ, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τις ευθύνες που φέρουμε και την ε, ανάγκη για κοινή προσπάθεια, για συνεργασία στο πρόβλημα αυτό. Όπως και με τη χρηματοπιστωτική κρίση. Είδαμε ότι υπάρχουν χώρες μέλη που αμφισβητούν ε, τις ε, δεσμεύσεις ως προς την υπεράκτια ανάπτυξη και ακόμη και το ποσοστό του 4% επί του ΑΕΠ και λένε ότι δεν χρειάζεται να προσφερθούν επιπλέον κονδύλια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Άρα, είτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, είτε άλλα κράτη στον κόσμο πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά με σοβαρότητα και αμέσως, γιατί εδώ δεν κρίνεται η τύχη της επόμενης γενιάς, κρίνεται η τύχη και η επιβίωση αυτής της δική μας γενιάς, το κατά πόσον θα επιβιώσουν τα νησιά σας τώρα. Και άρα η δική σας παρουσία, προετοιμασία, τα όσα έχετε να, μας πείτε είναι πολύ ευπρόσδεκτα εδώ. Η κλιματική αλλαγή, τα όσα έχετε να μας πείτε φυσικά ε, για, τις, για τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής έρχονται την στιγμή όπου βλέπουμε την υλοποίηση των κινδύνων και πιστεύω ότι θα δεχθείτε από πλευράς της πολιτικής μου ομάδα Σοσιαλδημοκρατών ότι δεν σας αφήνουμε να αγωνιστείτε μόνος σας και ότι αγωνιζόμαστε μαζί σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρνας έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Ήταν σαφής η παρουσίασή του και μας απέδειξε ότι θα πρέπει να χωριστούμε σε όλα τα μέτωπα ταυτόχρονα. Έχετε βέβαια να αντιμετωπίσετε τις ε, κλιματικές αλλαγές και αυτό σημαίνει πολλές ε, αλλαγές ως προς την συμπεριφορά, τη στάση των ανθρώπων στη χώρα σας. Μιλήσατε για, το, για την ανάγκη να μην αυξηθεί η θερμοκρασία κατά περισσότερο από 1,5 βαθμούς. Αγώνα σε όλα τα μέτωπα σημαίνει ταυτόχρονα αγώνα σε όλα τα μέτωπα και ω προ τη χρηματοδότηση. Και εσεί αναφερθήκατε στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη στην ομιλία σα. Θα πρέπει, πιστεύω, να καταστεί απόλυτα σαφέ στην Κοπενχάγη το κατά πόσον τα χρήματα που θα ζητηθούν, θα ζητηθούν να διατεθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στις αναπτυσσόμενες χώρες θα είναι συμπληρωματικά κονδύλια πέραν της δημόσιας ενίσχυσης προσφέρεται για την ανάπτυξη, όπως πιστεύω εγώ, ή εάν θα είναι χρήματα τα οποία θα αντληθούν από κάποιες δέσμες μέτρων ήδη αφιερωμένες στην ε, ε, αναπτυξιακή βοήθεια. Πράγμα το οποίο βέβαια θα σήμαινε υποβάθμιση της συνολικής ενίσχυσης για την ανάπτυξη και διαφορετικό χαρακτηρισμό της μόνο. Τα χρήματα που έχουμε τώρα στη θέση μας για την ανάπτυξη δεν επαρκούν ούτε καν για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας. Εσείς στην Κοπενχάγη εκφράσατε αυτές σας τις θέσεις, εξηγήσατε την κατάσταση και συμφωνείτε με αυτά τα οποία είπα εγώ. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ κύριε Πάνκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να πάρω το λόγο σήμερα το πρωί, γιατί σήμερα το πρωί ακριβώς δύο φορές αναφερθήκαμε σε δύο προβλήματα, σε δύο συνέπειες των κλιματικών αλλαγών. Πρώτα απ' όλα μιλήσαμε για τον Μπαγκλαντές, που εσείς ο ίδιος πρόεδρε παρουσιάσατε τη σχετική ε, κατάσταση και σήμερα το πρωί ακριβώς έμαθα ότι το λιώσιμο των παγετών στα Εμαλάγια οφείλονται στις κλιματικές αλλαγές, οπότε και το Μπαγκλαντές αναγκάζεται να πάρει μέτρα, για παράδειγμα να ανυψώσει χωριά για να μην πλημμυρίσουν από το νερό. Οι συνάδελφοι λοιπόν από τον Ειρηνικό που είναι εδώ, ο Πρωθυπουργό, πρέπει να τα ακούσει και πρέπει επίσης να ξέρει πως η δικιά του η φωνή όταν μιλάει για το τουβαλού που εγώ γνωρίζω πολύ καλά και όταν μιλάει για την άνοδο των υδάτων ε, γύρω από το νησί ε, ότι είναι και αυτό φαινόμενο που οφείλεται στις κλιματικές αλλαγές. Το τουβαλού λοιπόν πλημμυρίζει όταν έχουμε πλημμυρίδα, ε, η παλήρια δηλαδή είναι κάτι από το οποίο κινδυνεύει το Τουβαλού. Υπάρχει το Τουβαλού, υπάρχουν και άλλα μικρά νησιά που βρίσκονται πολύ κοντά σε εμά και που είναι αντιμέτωπα με τις κλιματικές αλλαγές. Συνεπώς, συμφωνώ με τα όσα μας είπε ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί και όντως πιστεύω ότι πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε το κοινοβούλιο μας σε αυτό το πρόβλημα. Είναι πρόβλημα που εμεί μπορεί να μην το ζούμε καθημερινά, αλλά οι άνθρωποι αυτοί το ζούνε στον ειρηνικό. Αν λοιπόν δεν φροντίσουμε να έχουν μέσα στη διάθεσή τους για να ανυψώσουν τη γη τους, να φτιάξουν φράγματα, προκειμένου να αποφευθούν οι πλημμύρες, ο κόσμος θα φεύγει, θα πηγαίνει σε άλλες υπήρους και θα το νιώσουμε αυτό και εδώ. Ένα εκατομμύριο από τον Παγκλαντές ακούσαμε σήμερα το πρωί ότι θα πρέπει να φύγουν και να έρθουν στις δικές μας χώρες. Συμφωνώ λοιπόν με τόσα μας είπε ο Πρωθυπουργό. Πρέπει να βρεθούν μέσα για να μην φεύγει ο πληθυσμός από εκεί. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Uh, thank you, Mr. Madam Levin. Ε, παρακαλώ, κυρία Λεβίν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ, που ήρθατε. Χάρηκα που σας άκουσα. Χάρηκα επίσης που σας άκουσα να λέτε ότι πρέπει να περιορίσουμε σε 1,5 την αύξηση της θερμοκρασίας και όχι σε δύο βαθμούς όπως έχουν συμφωνήσει οι ηγέτες. Βρίσκω αρκετά θαραλέο το να το λέτε. Όμως η απειλή με την οποία είμαστε αντιμέτωποι είναι τεράστια. Οι κλιματικές αλλαγές, πρέπει να ξέρουμε, δεν θα συμβούν σιγά σιγά. Είμαστε υπό την απειλή και ξαφνικών αλλαγών και μπορεί οι δύο βαθμοί να είναι πάρα πολύ για τον πλανήτη μας. Αν επιταχυνθεί επίσης η άνοδος της θερμοκρασίας στον πλανήτη μας, και αυτό μπορεί να δημιουργήσει απότομες αλλαγές λόγω των μηχανισμών που διέπουν το οικοσύστημά μας και έτσι μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με πολύ απότομες αλλαγές και καταστροφές για τις οποίες ο κόσμος να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε και αυτό που χρειάζεται σε όλους μας είναι να αλλάξουμε την νοτροπία όσον αφορά τις κοινωνίες μας. Μπορεί να ακούγεται ηρωνικό, αλλά υπάρχει κάτι που λέγεται The Happy Planet Index. Δηλαδή ο δείκτης του χαρούμενου πλανήτη. Είναι μια οργάνωση που προσπαθεί να εντοπίσει τι θέλει ο κόσμος, τι θέλουν οι κάτοικοι του βελού. Προσπαθούν να υπολογίσουν να δούνε δηλαδή πότε ένας άνθρωπος νιώθει χαρούμενος, με πόσους φυσικούς πόρους γίνεται αυτό, πόσο μπορείτε να προστατεύσετε τη φύση, την μητέρα γη, όντας ευχαριστημένη. Εσείς έχετε υψηλά επίπεδα ζωής και μια αντίληψη ευτυχίας η οποία συνάδει με την προστασία της φύσης. Έχετε λοιπόν εσείς πολλά να διδάξετε εμάς στις δυτικές χώρες και τους ηγέτες μας προκειμένου να αλλάξουμε νοτροπία για το τι θεωρούμε καλά στάνταρτ ζωής. Χαίρομαι και ελπίζω να μπορέσετε να τα πείτε αυτά και στην Κοπεχάγη σύντομα. Ευχαριστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διευθυντής Ρέιρα. Παρακαλώ. Πείτε μας, τι εννοούσατε με αυτά που ακούσαμε νωρίτερα. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε και εμείς σε αυτήν τη συζήτηση. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον Πρωθυπουργό του Τουβάλου που ήρθε εδώ σήμερα. Συμφωνούμε και εμείς με τις ανησυχίες που εξέφρασε όσον αφορά τα νησιά του Ειρηνικού. Δεν μιλάμε μόνο για κλιματικές αλλαγές, μιλάμε για την επιβίωση ορισμένων χωρών εκεί και για την ζωή χιλιάδων ανθρώπων. Συμφωνούμε με τις δράσεις που μας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Εμείς στις δράσεις μας όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία και τις κλιματικές αλλαγές πάντα ξεκινάμε από την αρχή που λέει ότι αυτοί που θα υποφέρουν περισσότερο είναι εκείνοι που συνεισφέρουν λιγότερο στο πρόβλημα, που δημιουργούν λιγότερο το πρόβλημα. Και γι' αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει εμείς να είμαστε πιο αυστηροί με τους εαυτούς μας και να στηρίξουμε την διαδικασία που έχει ξεκινήσει σε διάφορες αναπτυσσόμενες χώρες. Εμείς έχουμε ευθυγραμμιστεί με τους μηχανισμούς μας όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, όχι μόνο με αυτό που έχουμε ακούσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πάντως φροντίζουμε και για την ηθική στήριξη αλλά και για την οικονομική στήριξη. Και αυτό όχι μόνο για όλες τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά κυρίως ε, φροντίζουμε για τις λιγότερο προηγμένες χώρες. LDCs. Αυτό είναι θέμα επιβίωσης για αυτές. Επιτρέψτε μου να σας συγχαρώ για τις προσπάθειες που κάνετε στη χώρα σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Συχνά, σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες βλέπουμε ότι τα εθνικά τους προγράμματα προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές αποτελούνται από προγράμματα τα οποία μοιάζουν με τα στολίδια που βάζουμε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τα Χριστούγεννα. Χωρίς να έχουν πραγματική ουσία. Στην περίπτωση όμως του Ντουβάλου Στα πλαίσια της συνεργασίας μεταξύ μας μιλάμε για μια στρατηγική που έχει πολύ καλά σχεδιαστεί. Άρα ε, θα υπάρξουν καρποί από αυτή τη συνεργασία. Αυτή τη διαδικασία θα θέλαμε να τη βλέπουμε πιο συχνά και σε άλλες χώρες. Τώρα για να έρθω στα πιο συγκεκριμένα ζητήματα, κύριε Πρωθυπουργέ. Ξέρετε ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία μέσω του ενδεικτικού εθνικού προγράμματος και εσείς φροντίσατε να επικεντρωθεί η αναπτυξιακή μας συνεργασία σε θέματα νερού και υγιεινής. Χάρη λοιπόν στη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές, τη Συμμαχία για τις Κλιματικές Αλλαγές, πέρα από τα προγράμματα τα οποία θα στηριχθούν στα πλαίσια του φόρου για τις Μαλδίβες, για παράδειγμα, σκοπεύουμε με τα κονδύλια για το 2010 που ενισχύονται χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα φροντίσουμε λοιπόν να ε, βοηθήσουμε και το Τουβάλου. Θα ξεκινήσουμε συζητήσεις μαζί σας για να δούμε ακριβώς πώς θα μπορέσουμε να διαρθρώσουμε καλύτερα ε, την βοήθεια αυτή. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη την ιδέα σας για ένα trust fund. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ καλή ιδέα γιατί θα μας βοηθήσει να συγκεντρώσουμε τους πόρους που έρχονται από διάφορες πηγές. Στις συζητήσεις μαζί σας κύριε Πρωθυπουργέ πρέπει να εξετάσουμε αυτή τη δυνατότητα η οποία πιστεύω ότι πολλά έχει να προσφέρει. Είναι πραγματικά ο καλύτερος τρόπος για να ευθυγραμμιστούμε όλοι ε, στις δικές σας ανάγκες και στη δικιά σας στρατηγική. Πέρα αυτών, πρέπει να πω ότι ιδιαίτερα στον ειρηνικό οι κλιματικές αλλαγές δεν είναι εθνικό πρόβλημα, είναι περιφερειακό Έτσι λοιπόν στα πλαίσια του ενδοακέ οικονομικού πακέτου θέλουμε να στηρίξουμε και περιφερειακές οργανώσεις που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές αλλαγές. Έτσι έχουμε βάλει 8 εκατομμύριο ευρώ για ολόκληρο τον ειρηνικό προκειμένου να αντιμετωπιστούν κλιματικές αλλαγές. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να εξετάσουμε και τη δυνατότητα τα κονδύλια αυτά να πάνε και μέσω στήριξη στον προπολογισμό όπου γίνεται, ώστε να δοθούν προκαταβολές και να επιταχυνθεί η εφαρμογή των προγραμμάτων. Επιπλέον, θα έχουμε και άλλα 8 εκατομμύρια αποκλειστικά για μικρές ε, χώρες νησιά του Ειρηνικού. Συνεπώς έχουμε μια καλή στρατηγική που μας επιτρέπει να ενισχύσουμε την συνεργασία. Προστακούμε επιπλέον συζητήσεις μαζί σας κύριε Πρωθυπουργέ, ώστε τα πράγματα να ξεκινήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πάντως για άλλη μια φορά και χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Συμμαχία για τις Παγκόσμιες Κλιματικές Αλλαγές μας βοηθάει να επιταχύνουμε τον πολιτικό διάλογο με τις χώρες ΑΚΕ και τις υπονάπτυξη χώρες. Με πειραματικά προγράμματα πάντως στην περίπτωση του Τουβάλου περιμένουμε ότι θα έχουμε καρπούς πολύ γρήγορα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Διευθυνταρέρα. 8 εκατομμύρια είναι για πειραματικά προγράμματα. Και αν πάνε καλά, τότε θα υπάρξει περισσότερη, περισσότερα κονδύλια, μεγαλύτερη χρηματοδότηση. Έτσι δεν είναι, ο κύριο Ρέιρα. καλά προσπαθείτε, αλλά good try. Αλλά θα εξαρτηθεί. Θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της Κοπεχάγης και την δημοσιονομική αρχιτεκτονική που θα έχουμε μετά. Σε αυτό το στάδιο πρόκειται για κονδύλια τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας για να ξεκινήσει η περιφερειακή αυτή διάσταση αντιμετώπιση των ειρηνικών των κλιματικών αλλαγών. Ε, σίγουρα ανάλογα με τα αποτελέσματα. Πάντως ένα από τα σημεία κλειδί εδώ για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών είναι να ε, μας υποβάλλονται καλές στρατηγικές. Ειλικρινά πιστεύω ότι μέσω πρόθεσμα, αν οι στρατηγικές υπάρχουν, πάντα ανάλογα με τα αποτελέσματα της Κοπεχάγης, έτσι, πάντως θα ακολουθήσουν και κονδύλια. Και όχι μόνο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από άλλες πλευρές. Εδώ μιλάμε για μια περίπτωση που έχουμε μια πολύ καλή στρατηγική δεν είναι ότι προσπαθούμε από δεξιά και αριστερά έτσι να βρούμε λεφτά χωρίς να υπάρχει μια καλή ε, στρατηγική. Την έχουμε την καλή στρατηγική. Οπότε θα στηρίξουμε τέτοιες περιπτώσεις. Ευχαριστούμε κύριε Ρέρα. Δεν ξέρω αν ήσασταν εδώ όταν συζητάχαμε για κλιματικές αλλαγές νωρίτερα. Ο συνάδελφός σας ήταν εδώ. Και αναφέρθηκε και στα Ηνωμένα Έθνη. Την έκθεση Ουρτάνιο Λέντε που λέει ότι αν έχουμε προσαρμογές καλές στις κλιματικές αλλαγές, ε, μπορούμε να επιταχύνουμε και την ανάπτυξη. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Αν πάνε κονδύλια στις κλιματικές αλλαγές για την καταπολέμηση κλιματικών αλλαγών, συγχρόνως επιταχύνεται και η ανάπτυξη. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχετε κονδύλια EDF, συνεπώς οι προσαρμογές στις κλιματικές αλλαγές θα μπορούσαν να αποτελέσουν και μία mainstream δραστηριότητα για την ανάπτυξη. Σωστά. Ναι, ναι, ασφαλώς. Δεν θέλω να αρχίσω να φιλοσοφώ εδώ, αλλά πιστεύω ότι ο προβληματισμός μας για τις κλιματικές αλλαγές ε, σιγά σιγά αλλάζει και την αναπτυξιακή νοοτροπία. Και πέρα από τη χρηματοδότηση κάποιων προγραμμάτων <clears throat> κατά των κλιματικών αλλαγών, όντως αλλάζει συγχρόνως συνολικά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριος Γκουτζάντς. Παρ' όλα αυτά παραμένει το εξή ερώτημα. Αν πάρουμε από τα κονδύλια που είναι για τη δημόσια στήριξη και τα πάμε στι κλιματικέ αλλαγές, τι θα γίνει. Εδώ θέλει η Κομισιόν να μου τα πει ξεκάθαρα. Υπάρχουν χώρε οι οποίε συμφωνούν με μένα και άλλε που έχουν την αντίθετη άποψη. Γι' αυτό και η Ευρώπη καλά θα κάνει να ξεκαθαρίσει τη θέση τη πριν πάει στην Κοπεχάγη να τα πει. Είναι πολύ σημαντικό. Αν θέλουμε συμφωνία θα πρέπει να έχουμε μια διπλή πλειοψηφία και όλων των χωρών και των χωρών του παραρτήματος 1 που είναι υπεύθυνε για την ρήπανση. Διπλή πλειοψηφία λοιπόν πρέπει να υπάρχει. Και αν θέλουμε να δούμε πρώτα τι υπονάπτυξη χώρε, η Ευρώπη δεν θα πρέπει να αφήσει καμία αμφισημία. Αλλιώ θα είμαστε υπεύθυνοι για ένα συλλογικό ψεύδος. Δεν ξέρω ο κύριος Ρέιραν θέλει να απαντήσει. Είναι σαφές ότι δεν θα πρέπει να σταματήσουμε τα προγράμματα που είναι ήδη εν εξελίξη. Γιατί έχουμε προβλήματα με τη χρηματοδότηση της καταπολέμησης των κλιματικών επιπτώσεων. Οποιαδήποτε χρηματοδότηση σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να σημαίνει μείωση της ε, στήριξης και της χρηματοδότησης των υπαρχών των προγραμμάτων. Άκουσα τον Πρωθυπουργό του Τουβαλού στη Στοκχόλμη τη μέρα της ανάπτυξης. Εσείς ήσασταν. Εσείς δεν το είπατε. Α, όχι, το ήταν κάποιος άλλος συμπολίτης σας, κάποιος άλλος από τον Τουβαλού. Είμαι σίγουρος ότι αυτά που θα πω τα είπε κάποιος από τον Τουβαλού. Σας είπε και είπατε ότι η χώρα σας βυθίζεται. Στην Κοπεχάγη σήμερα υπάρχουν φήμες ότι κάποια ευρωπαϊκά κράτη λένε πως κάποια από τα μέτρα θα μπορούσαν να πληρωθούν από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια για την καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή. Διαφωνώ με τον κύριο Γκέρνη ότι αυτό είναι απαράδεκτο. Γιατί η χρηματοδότηση των μέτρων προσαρμογή, μετριασμού των επιπτώσεων είναι μια προπόθεση για να υπάρξει ανάπτυξη αδιανόητο για μένα, για τους συναδέλφους, να χρηματοδοτήσουμε από την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια τα μέτρα τα οποία πρέπει να χρηματοδοτήσουμε. Ε, είμαστε δεσμευμένοι, εμείς είμαστε υπόχρεοι. Είναι η εφαρμογή της αρχής του ορυπαίνου πληρώτη και ελπίζω ότι θα υπάρχει πληροψηφία εδώ για να σταματήσουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι πραγματικά αυστηρή σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, Ξέρω ότι έχετε πολλές ανηλυμένες υποχρεώσεις. Βλέπετε όμως ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Ίσως θα θέλατε λοιπόν να πείτε κι εσείς λίγα λόγια εν είδη απάντησης. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι βουλευτές, Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για τη συνεισφορά σας. Ήταν πολύ ενημερωτικά όλα αυτά που είπατε. Θεωρούμε ότι είναι η ένδειξη της δέσμευσης που έχετε αναλάβει. Ε, και θεωρώ ότι η δέσμευση αυτή απέναντι στη χώρα μου και στις άλλες ευάλωτες χώρες με... για μια χρηματοδότηση από... Η δέσμευση αυτή είναι ικανοποιητική από πλευρά σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό το μέσο χρηματοδότησης για τα προγράμματα νερού στη χώρα μου. Αν κατάλαβα καλά, η χρηματοδότηση θα ξεκινήσει κάποια στιγμή μέσα στο 2010. Θα ήθελα να ξεκινήσει η χρηματοδότηση το συντομότερο δυνατόν, ούτως ώστε να βοηθηθεί ο πληθυσμό μας. Και όπως είπε και ο εκπρόσωπος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, οι επιπτώσεις γίνονται αισθητέ ήδη σήμερα. Δεν θα γίνουν αύριο μεθαύριο. Θα θέλαμε λοιπόν η βοήθεια αυτή να δοθεί το συντομότερο δυνατόν. Ε, Τώρα, αυτό πρότεινε ο κύριος Κάσμαν. Αν θα πρέπει δηλαδή η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια να διαιρεθεί. Ε, ένα τμήμα να πάει για την ε, προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές. Εμείς θα θέλαμε νέα χρηματοδότηση αν η επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια διαιρεθεί, νομίζω τότε θα διασαλευθεί η αναπτυξιακή μας πορεία. Αν ένα τμήμα δηλαδή αυτής της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας πάει σε μέτρα προσαρμογής ε, στις κλιματικές αλλαγές. Σας ευχαριστώ όλοι και ο κύριος Ντέβα και εγώ που μπορέσατε να έρθετε και ελπίζω να έχουν αρθεί οι όποιες απορίες υπήρχαν ε, από την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, θέλω να το πω επίσημα τώρα ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, καμία παρεξήγηση α, σε σχέση με αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στη συνομιλία στην Κοπενχάγη. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα είναι στο Στρασβούργο. Στις 14 μεταξύ 7 και 8.30 το βράδυ. Δευτέρα το πρωί. Δευτέρα το απόγευμα, συγγνώμη. Περιμένουμε την έγκριση της διάσκεψης των Προέδρων και θα κάνουμε και την 5η 17 Δεκεμβρίου 9 με 10.30 για να ε, συναντήσουμε τους ε, ε, ανθρώπους που πήραν φέτος το βραβείο Ζαχάροφ από τη Ρωσία. Είναι μια κοινή συνεδρίαση με την ΑΦΕΤ. Και στις 25 Ιανουαρίου, Δευτέρα, θα έχουμε την επόμενη συνεδρίασή μας στις Βρυξέλλες. Αυτά ευχαριστώ.